Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, προτείνω να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουμε καταρχήν την ώρα των ερωτήσεων προς την Κομισιόν ως πρώτο σημείο στην μέση διάταξη της δεύτερης μέρας συνεδρίασής μας. Η πρότασή μου είναι να προχωρήσουμε προς το σημείο υπαριθμών 6 και να ζητήσουμε τον κύριο Ντόρσκης να παρουσιάσει το ερώτημα του προς την Κομισιόν. Αυτοί οι οποίοι μας ακούνε βέβαια πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς συζητάμε. Μπορείτε να εξηγήσετε το ερώτημά σας και μετά να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Κύριε Ντόνσκης, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Να το περιγράψω εν συντομία. Η ουσία του ερωτήματος είναι ότι μέχρι τώρα η Κίνα εμπόδιζε συστηματικά όλες τις πρωτοβουλίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις προσπαθίες μας να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας <clears throat> για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώ στην ίδια πορεία, αλλά μπλοκάρουν όλε τι πρωτοβουλίε μα οι Κινέζοι. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχει κάτι καινούριο σε επίπεδο εργαλείων που οι μέσων θα μα δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Ντόνσκι. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. είναι κάπως διαφορετικό το ερώτημα από το γραπτό ερώτημα του κύριου Ντόνσκης. Εάν μου επιτρέπετε θα απαντήσω πρώτα στο γραπτό ερώτημα και μετά θα κάνω ένα πιο γενικό σχόλιο για το Θιβέτ. Είναι σαφές ότι έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, σημαντικά διαφορετικές προσεγγίσεις για το θέμα του Θιβέτ από ότι η Κίνα. Εμείς ανησυχούμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και για το γεγονός ότι η πρόσβαση στο Θιβέτ για τα διεθνή μέσα ενημέρωση τους διπλωμάτες και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και παραμένει περιορισμένη. Εξάλλου δεν υπήλθε μεγάλη πρόοδος στις επαφές μεταξύ Δαλάη Λάμα και κινέζικων αρχών. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Θιβέτ δεν αφήνει περιθώριο αμφισημίας και παρανοήσεως. Έχει τονιστεί πολλές φορές στην ε, Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει εκφραστεί με τα ψηφίσματά του. Και θέλω να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα της Κίνας που περιλαμβάνει και το Θιβέτ. Δεύτερον, υποστηρίζουμε πάντα την ειρηνική συμφιλίωση μέσω διαλόγου μεταξύ Κινέζικων Αρχών και εκπροσώπων του Δαλάη Λάμα. Τρίτον, πιστεύουμε ότι ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι επικοδομητικός και ουσιαστικός. Να αντιμετωπίσει όλα τα βασικά θέματα, <clears throat> όπως είναι η διατήρηση της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Θιβέτ, της θρησκευτική και πολιτιστικής του παράδοσης και της επίτευξης ενός λογικού συστήματο αυτονομία στο Θιβέτ. Και επίση θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των Θιβέτιανών στη λήψη απόφαση. Για μα, λοιπόν το Θιβέτ είναι ένα θέμα κυρίω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε μεταδώσει αυτό το μήνυμα κατά επανάληψη και κατά συρροή στου Κινέζου ομολόγου μα και έχουμε κάνει σαφέ ότι αυτή είναι η απόψη μα. Κάνουμε κάθε προσπάθεια να κατανοήσουμε τη θέση του σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Αλλά συμφωνούμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και η κατάσταση στο Θιβέτ είναι πηγή θεμητής ανησυχίας για την διεθνή κοινότητα, κάτι το οποίο τονίσουμε στους Κινέζους συνομιλητές μας, είτε στα πλαίσια του διμερούς διαλόγου ανθρωπινών δικαιωμάτων, κάθε φορά λοιπόν το εγείρουμε αυτό το θέμα, και επίσης και στην, στα πλαίσια της πρόσφατης αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Θιβέτ, γιατί όπως ξέρετε η Κομισιόν έχει ήδη πληροφορήσει την ε, υποεπιτροπή σας σε μια και κλεισμένο των θυρών συνάντηση για αυτή την αποστολή. Για τον Κινέζικο-Θιβετιανό διάλογο τώρα. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Θιβετιανή πλευρά έχει επαναλάβει την ε, ρητή της δέσμευση να μην αναζητήσει, να μην επιζητήσει την ανεξαρτησία και χαιρόμαστε που ακολουθεί τον μέσο δρόμο ο Δαλάη Λάμα για μια αποδεκτή αμοιβαία και μόνιμη λύση. Για το ερώτημα του κυρίου Ντόνσκης για το θέμα της ε, παρουσίας ενός του διορισμού ενός ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Θιβέτ. Εγώ θα πρέπει να εκφράσω αμφιβολίες για το αν θα προκύψει προσθέμενη αξία από το διορισμό ενός τέτοιου αντιπροσώπου όταν ήδη υπάρχουν σημαντικοί τακτική διάβλη επικοινωνία, κυρίω μέσα στα πλαίσια του διμερού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι ένα τέτοιο απεσταλμένο δεν θα έχει δυνατότητα να παίξει ένα αποτελεσματικό ρόλο λόγω εμποδίων που θα θέσει η Κίνα, γιατί η Κίνα δεν θέλει καμία μορφή διεθνού διαμεσολάβηση για το Θιβέτ. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Απεσταλμένος ποτέ δεν έχει πατήσει το πόδι του στο Θιβέτ. Γιατί τον εμπόδισαν οι κινέζικες αρχές. Επομένως, εμείς χαιρετίζουμε ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επαφές τους παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρούμε απτά αποτελέσματα. Για το Θιβέτ, λοιπόν, εμείς έχουμε εκφράσει σαφώς τις ανησυχίες μας και τις επιθυμίε μας και ξέρουμε και έχουμε αναφέρει πάντα το πώς έχει επηρεάσει η κινέζικη παρουσία στον τρόπο ζωής του Θιβέτ. Έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας επίσης για το γεγονός ότι όλοι οι νομάδες και κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εγκατασταθούν σε μόνιμα συμπλέγματα κατοικιών. Και αυτό θα έχει προφανές, προφανή αντίκτυπο στον παραδοσιακό του τρόπο ζωής. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο συζητούμε κάθε φορά με τους Κινέζους συνομιλητές μας. Εξάλλου όμω, ο διάλογο είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει άλλο ένα γύρο διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλο του έτου και επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή πλήρω. Τελευταίο και λουκούμιο σημείο για το τι μπορούμε να κάνουμε για την Κίνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αυτό είναι μια συνεχιζόμενη και ευρεία συζήτηση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπίστηκαν στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, όπου έγινε σαφές από τη δική μας πλευρά ότι είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας εταιρική σχέση με τους Κινέζους στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς κάνουμε πάντα μια πάρα πολύ στεναρή έκκληση να μπορέσει να γίνει σεβαστή η Διεθνή Σύμβαση για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα. Το εργαλείο μας λοιπόν είναι ο διμερής διάλογος και πάντα αντανακλώμε και απηχούμε τις ανησυχίες σας στους Κινέζους και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε, να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποσχεθήκατε ότι θα μας δώσετε κάποιες συμπληρωματικές απαντήσεις στη ερώτημα του κυρίου και αν υπάρχουν νέα μέσα ή το καλύψατε και αυτό. Θέλετε να συνεχίσετε, συνάδελφε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την απάντηση και τα σχόλιά του. Αλλά σχετικά με το Θιβέτ νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει διότι αφενός μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για στρατηγικές και κατακαιρματισμένες οι οποίες ε, να καλύπτονται από επιμέρους μέσα αλλά χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο Θιβέτ και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μέσα. Γι' αυτό παροτρύνω τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στις 6 Δεκεμβρίου στη συνεδρίασή μας σε αυτό το θέμα όταν θα συζητήσουμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Το αφήνουμε λοιπόν κατά μέρος επί του παρόντος. Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας. Το επόμενο, η επόμενη ερώτηση, Μπάρμπαρα Λόχβιερτ, υπαριθμών 3. Μπορείτε σύντομα να μας παρουσιάσετε το περιεχόμενο της ερώτησής σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε αφορά την ελευθερία του τύπου στην Ταϊλάνδη. Η κατάσταση επιδεινώνεται σύμφωνα με τους ε, reporters χωρίς σύνορα. Στο Press Index Worldwide έχει, κατέχει τα Ιρλανδία θέση 113, ενώ ήταν στο 65 προηγουμένως. Η ερώτησή μου σχετίζεται με αυτό. Ερωτώ την Επιτροπή ποια είναι η αξιολόγησή της σχετικά με την ελευθεροτυπία στην Ταϊλάνδη. Και επίσης αναφέρομαι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, την κυρία Σινανού Πενκόν, η οποία είναι η εκδότρια της ε, εφημερίδας Ιντερνετ αλλά συνελήφθη για δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο, ε, όταν γύριζε, επέστρεφε από μια διάσκεψη για την ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία. Η ερώτηση είναι κατά πόσον παρακολουθεί τη δίκη εναντίον της Επιτροπή και το, το έχει περιλάβει αυτό το θέμα σε συναντήση με την Ταϊλανδέζικη κυβέρνηση. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωβουλευτή που έθεσε αυτό το ερώτημα. Για την πρώτη ερώτησή σας λοιπόν, σχετικά με την αξιολόγηση της ελευθεροτυπίας στην Ταϊλάνδη από την Κομισιό, το το διάταγμα του Απριλίου εξακολουθεί να ισχύει σε τέσσερις επαρχίες συμπεριλαμβανομένες και την Μπαγκόκ, της πρωτεύουσας. Επίσης υπάρχουν πολύ σημαντικοί περιορισμοί στην ελευθερία του τύπου. Μέσα ενημέρωσης τα οποία υποστηρίζουν την αντιπολίτευση επίσημα, επίσημα στοιχεία ε, των μέσων ενημέρωσης που έκλεισαν μετά από αυτό το διάταγμα δεν είναι απόλυτα σαφή. Μια καλωδιακή τηλεόραση, People Channel, το κανάλι του λαού και άλλες εφημερίδες που των ε, ρηθρών, των Reds, UDD έχουν, αναγκάστηκαν να κλείσουν. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί επίσης δεν τους επιτρέπεται να λειτουργούν πλέον. Τους αφαιρέθηκε η άδειά τους και 49 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί. Τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης έχουν επηρεαστεί από τη λογοκρισία της κυβέρνησης η χώρα αναφερόταν σε ε, μια χώρα υπό εποπτεία, υπό επιτήρηση στην έκθεση Enemy on the Internet στις 11 Μαρτίου 2010 ανακοινώθηκε αυτό από τους ρεπόρτες χωρίς σύνερα. Η εφαρμογή, η εφαρμογή του νόμου για την λειτουργία του διαδικτύου μετά από εντολή του δικαστηρίου αυξήθηκε από δύο περιπτώσεις το 2007 σε 42.660 περιπτώσεις την περίοδο από Ιανουάριο μέχρι Σεπτέμβριο 2010. Το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης περιορίζεται από την κατάσταση κατεπίγοντος που ανακηρύχθηκε στις 7 Απριλίου και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Μάιο και τον Απρίλιο 2010 στην Μπαγκόκ. Το διάταγμα επιτρέπει στις αρχές να διακόπτουν τη λειτουργία ιστοσελίδων χωρίς δικαστική εντολή και αυτό αφορά παραπάνω από 100.000 περιπτώσεις. Μιλάμε λοιπόν για ανησυχητική κατάσταση. Ο Πρωθυπουργό το Δεκέμβριο του 2009 παραδέχθηκε ότι υπήρχαν προβλήματα με την εφαρμογή αυτού του νόμου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά η κυβέρνησή του δεν φαίνεται να, λαμβάνει, ε, είναι, να επιδεικνύει οποιαδήποτε ευαισθησία σε ό,τι αφορά την παρενόχληση των μέσων ενημέρωσης. Το Υπουργικό Συμβούλιο τον 15 Ιουνίου του 2010 δημιούργησε ένα γραφείο πρόληψης και κατάργησης των εγκλημάτων ε, που έχουν σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ε, δήθεν με σκοπό να προστατεύσει τη βασιλική οικογένεια. Σχετικά με τη δεύτερη ερώτησή σας για την κατά πόσο παρακολουθεί την ε, δίκη της Ιρανούκ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά πόσο έχει θέσει αυτό το θέμα στις συναντήσεις της με την Ταϊλανδέζικη κυβέρνηση, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρακολουθεί την, τα θέματα της ελευθεροτυπίας και της εξελίξης σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στην περίπτωση του Ιρανούκ, ειδικότερα στην Ταϊλάνδη ο πολιτικός σύμβουλος συναντήθηκε με την ίδια τη Ιρανούκ στην Μπαγκόκ μετά την απελευθέρωσή της με εγγύηση και άκουσε τις ανησυχίες που διατύπωσε. Μια, ένα δελτίο τύπου ετοιμάζεται από τον πολιτικό σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μπαγκόκ αναλύοντας το θέμα με σκοπό να να ενισχυθούν οι πολιτικές παρεμβάσεις. Στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κουνκάν, η περίπτωση της Ιρανούκ ειδικότερα συζητήθηκε συγκεκριμένα με τον ίδιο τον κυβερνήτη και τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές αρχές που βρίσκονταν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη δίκη η οποία πρόκειται να λάβει χώρα το Φεβρουάριο του 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθεί να υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθεροτυπίας γενικά και της περίπτωση της Ιρανού ειδικότερα στις τακτικές επαφές με τις ταλλανδέζικες αρχές, επίσης στο πλαίσιο των συναντήσεων υψηλού επίπεδου υψηλού επίπεδου που έγινε στα περιθώρια της ΑΣΕΜ στις Βρυξέλλες στις αρχές του Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Βαν Ρομπέγ, ανέφεραν τις ανησυχίες τους στη, στη συνάντηση με τον Ταϊλανδέζο ε, Ταϊλανδό Πρωθυπουργό, ανησυχίε που αφορούν την ελευθεροτυπία και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα στην Ταϊλάνδη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία μέσω της αντιπροσωπείας στην Ταϊλανδή για την παρακολούθηση αυτών των περιπτώσεων, για των περιπτώσεων παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την πολύ ολοκληρωμένη απάντηση και η οποία δείχνει και πάλι ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά στην Ταϊλάνδη και δεν ξέρω αν αυτή δεν είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν θέμα κατεπήγων. Πράγματι. Τώρα ερχόμαστε στην ερώτηση 1 του συναδέλφου Γκόλ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με δύο λόγια την ερώτηση και μετά θα μιλήσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αφορά έναν Ουιγούρο ε, πρόσφυγα. Ε, ε, του έχει δοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Ε, τώρα κινδυνεύει να εκδοθεί από τις καζακικές αρχές πίσω στην Κίνα ε, μετά από κινέζικες πιέσεις. Ε, γνωρίζουμε άλλες περιπτώσεις Ουιγούρων και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, η Κομισιόν να κινηθεί για αυτό το θέμα, να κάνει κάτι. Ευχαριστώ. Είναι μια πολύ σοβαρή ε, υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι την έχουμε ε, αντιμετωπίσει στέλνοντας μια επιστολή στον πρέσβη του Καζακστάν, η Κομισιόν. Η Κομισιόν παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην περίπτωση αυτή εδώ και πολλούς μήνες το άτομο αυτό ε, αναγνωρίστηκε ως πρόφυγας από, την, από το Γραφείο Προσφύγων του ΟΗΕ. Ε, έχει, του έχει αρνηθεί το Σεπτέμβριο από τις καζακικές αρχές το καθεστώς του πρόσφυγα. Το Γραφείο των Προσφύγων του ΟΗΕ έχει ειδική ευθύνη, είπα τη αρμοστία, έχει ειδική υποχρέωση να προστατεύσει το άτομο και να μην επιστραφεί το άτομο αυτό σε μια χώρα που μπορεί να βασανιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσεγγίσει τις κασικές, καζακικές αρχές και στις Βρυξέλλες και στην Αστάνα για να ε, πιέσει τις αρχές αυτές να εκδώσουν ε, τον, το άτομο αυτό, τον Ουιγούρο, προς ε, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. χθε είχαμε μία ακρόαση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, στο Καζακστάν η οποία έχει και την προεδρία της ΟΑΣΕ. Ε, καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν και ο πρόεδρος του Καζακστάν, ο κ. Ναζαρμπάιεφ, ε, επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ε, θα συναντήσει τον πρόεδρό μας και θα συζητηθούν διάφορα θέματα τα οποία συζητήσαμε και χθε στην ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Γκάλ. Έχετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση. Νομίζω ότι πρέπει το θέμα να παραμείνει ανοιχτό. Και κάθε φορά που υπάρχει ευκαιρία να θέτουμε αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω και στην συνάντηση που θα γίνει στο Καζακστάν ε, με μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, αυτά τα ανθρώπινα θέματα θα πρέπει να τα θέτουμε. Χθες ακούσαμε ότι οι καζακικές αρχές ε, κατάφεραν να ακυρώσουν την παράλληλη αυτή συνάντηση που θα γίνει με την Σύνοδο Κορυφής στην ε, Αστάνα. Είναι μια συνάντηση που προτίθενταν να οργανώσουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι αρχές της ΟΑΣΕ είναι ουσιαστικά συνεργασία με την ε, κοινωνία των πολιτών. Αυτό λοιπόν η στάση των καζακικών αρχών αγνοεί αυτή την αρχή. Τώρα μια ερώτηση δική μου για την χρηματοδότηση στην Τινησία και στην Αλγερία. Έχουμε εκθέσεις ότι η κοινωνία των πολιτών δεν έχει λάβει τη χρηματοδότηση αυτή. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν το νέο ποινικό κώδικα, το άρθρο 61α του ποινικού κώδικα που απαγορεύει οποιονδήποτε να πλήττει την οικονομική ασφάλεια της α, Ισίας. Ο υπεύθυνος υπουργός εξήγησε ότι το ε, ε, δίνει κίνητρα κάνει σε ε, να δίνει ας πούμε κίνητρα για να μην επενδύουν στην Τινησία σημαίνει ότι επιβουλεύεται τα συμφέροντα της Τινησίας. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και θα ήθελα να μας πει ο κ. Χέρτσοκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει ακριβώς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας. Προσπαθούμε να συζητήσουμε και με την Τινησία και με την Αλγερία το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιώντας τη Συμφωνία ε, Συνεργασίας και τον διαφθομένο διάλογο με την Τινησία. Είμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης των ε, διατάξεων ε, για τη συνεργασία αυτή. Για τη χρηματοδότηση τώρα η εικόνα είναι μεικτή. Στην Τινησία από το 2002 είχαμε τρία προγράμματα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ε, για θέματα φύλων, ε, για δημιουργία οργανώσεων προάσπισης των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία συνδικαλισμού, συνδικάτων. Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην Τινησία. Όπως αναφέρεται η κυρία Χαουτέλα, υπάρχει το νέο άρθρο 61α του ποινικού κώδικα που μπορεί όντως να έχει επιζήμιες επιπτώσεις, ε, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, αλλά ακόμα και πριν εισαχθεί αυτό το νέο άρθρο, αυτά τα προγράμματα αντιμετώπισαν δυσκολίες. Παραδείγματο χάρη, είχαμε ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρηματοδότηση ε, μπλοκαρίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Τινησίας. Οι αρχές θεωρούν ότι όλες οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να σταματήσουν ε, λόγω εσωτερικών προβλημάτων μέχρι να συνεδριάσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ήρθα σε επαφή με την Τινησιακή Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ενημερωθώ. Είναι ένα κλασικό πρόβλημα που έχουμε αυτό στις χώρες αυτές. Προς το παρόν Η προκήρυξη διαγωνισμού για προγράμματα για την, την Ισία δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες, γιατί η τοπική αντιπροσωπεία έχει εκτιμήσει ότι η κατάσταση εκεί δεν επιτρέπει την δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών στον τοπικό τύπο. και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων του μέσου εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία πέντε χρόνια διάφορες προτάσεις που λάβαμε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Τινησίας είναι περιορισμένος Υπάρχουν όμω κάποιες δραστηριότητε οι οποίες έχουν προχωρήσει και εφαρμόζονται τώρα. Φυσικά, όπου μπορούμε θα κάνουμε διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι τα προγράμματα αυτά θα εξαρτώνται και από την ε, ζήτηση. Σε ό,τι αφορά το 61α του ποινικού ε, κώδικα έχουμε επαφές με την, ε, μέσω της αντιπροσωπείας μας στην Τινησία και μέσω του Επιτρόπου Φιούλε για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων αυτών. Υπάρχει ένα επίσημο ανακοινωθέν που, από πλευράς της νησίας που, μας, που λέει ότι ο νόμος αυτός δεν περιορίζει την, τις δραστηριότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί ο τροποποιημένος νόμος Τώρα, για την Αλγερία. Από το 2002, 33 προγράμματα ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ ε, με 17 μικροπρογράμματα που εφαρμόζουν τοπικές οργανώσεις και δύο μεγάλα προγράμματα που εφαρμόζουν ε, οι διεθνείς οργανώσεις στην εργασία με τοπικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει. Και σε αυτά τα προγράμματα καλύπτουμε δικαιώματα παιδιών, καταπολέμηση της βίας στα σχολεία, ε, καταπολέμηση του AIDS, ε, δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού και οργανώσεων ε, κτλ. Καλύπτουμε πολλά θέματα. Υπάρχει συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις στην Αλγερία και αυτό το δείχνουν οι προκηρύξεις τοπικών διαγωνισμών και όλες οι δυνατότητες το 2008 και 2009 χρησιμοποιήθηκαν. Έχουμε και πολλές προτάσεις ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Ε, υπάρχουν και άλλα μέσα μέσω των οποίων χρηματοδοτούν τέτοια προγράμματα, μέσω φορέων και μέσω της πολιτικής γειτονίας επίσης. Um, Ευχαριστώ. Μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με το, την εφαρμογή του άρθρου 61α ε, στην Τινησία. Στην Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχετε διαπιστώσει και στους ίδιους ότι είχαμε ανταλλαγές απόψεων με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, οι οργανώσεις της Τινησίας ε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Έχουν φοβηθεί από αυτό το, νόμο. Ε, έχει δηλαδή ένα πολύ αρνητικό, μια πολύ αρνητική επίπτωση στην κοινωνία αυτό το άρθρο. Τώρα, να υπενθυμίσω σε όλους ότι η Υποεπιτροπή αποφάσισε πρόσφατα να στείλει μια αντιπροσωπεία στην Τινησία στις αρχές του 2011. Τώρα, λοιπόν, καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ετήσια έκθεση της ε, Αντιπροέδρου μας Λάιμα Αντρικίνε, που είναι η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Συγχαρητήρια αγαπητοί συνάδελφε. Έχετε προκαλέσει 423 τροπολογίες ε, στην έκθεσή σας, δηλαδή το έργο σας είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Εγώ στη δική μου ε, έκθεση είχα μόνο 200, τις μισές. Εσείς έχετε διπλάσια επιτυχία. Πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, πιστεύω ότι θα βρούμε τους αναγκαίους συμβιβασμούς, ούτως ώστε να στείλουμε ένα στεναρό μήνυμα πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ύπατο ε, εκπρόσωπο όταν γίνει η μεγάλη συζήτηση το Δεκέμβριο ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ολομέλεια. Ε, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου δηλαδή. Είναι μία από τις δύο μεγάλες ετήσιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τα θέματα που καλύπτουμε στο σχέδιο έκθεσης ε, μέσω των τροπολογιών φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο δίνει σημασία στο διάλογο για αυτά τα θέματα και πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια και πρέπει να βελτιωθούν και τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Αυτό το αναφέρουμε συστηματικά. Μιλάμε για την, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το τονίζουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα, την, την κατάστασή τους. Ε, υπάρχει και σχετικό ψήφισμα. Επίσης η θέση των γυναικών, η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία πεπιθήσεων. Υπάρχουν κάποιες νέες ενδιαφέρουσες προτάσεις και οι διεθνείς συμφωνίες για την εμπορική πολιτική καθώς ε, και οι ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις συμφωνίες. Ε, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ αυτό το θέμα γιατί έχουμε νέες αρμοδιότητες. Πολλές α, ε, χώρες κατονομάζονται. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά από την εισηγήτριά μας. Θα σχολιάσει η συγκήτρια της τροπολογίας και μετά θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ο Χάουιτ από τους σοσιαλιστές, Ντόνσκι από τους φιλελεύθερους, εγώ από τους πράσινους, ο Τάνοκ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές και Μπέρτσιεφ από την ΚΟΕ. Είναι οι σκιώδεις εισηγητές λοιπόν. Βεβαίω μπορεί να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, σήμερα είναι η δεύτερη εξέταση στην Υποεπιτροπή και θα το συζητήσει και θα ψηφίσει στις 9 Νοεμβρίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα το συζητήσει μετά η Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, στις 15 Δεκεμβρίου. Εισηγήτρια. Ευχαριστώ, λέει κυρία Ανδρίκηνα. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για την ιδιαίτερα ενεργή του συμμετοχή στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης που οδήγησαν σε 423 τροπολογίες. Επί τη βάση του έγγραφου εργασίας που συζητήσαμε πριν από μερικές Γνωρίζω ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για την κατάθεση τροπολογιών Παρά το γεγονός αυτό, ο αριθμός των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί με γεμίζει από αισιοδοξία. Και πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας αυτής, δηλαδή η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 θα είναι ο καρπός της κοινή μας εργασίας. Και θα αντανακλά τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σύνολη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε συμβαστικέ λύσει για τα κύρια επίμαχα θέματα, όπω είπα και προηγουμένω. Ο στόχο μου είναι να μπορέσω να έχω ένα όσο το δυνατόν πιο θετικό πνεύμα σε σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Οι πιο πολλές από αυτές τις τροπολογίες έχουν να κάνουν με το διεθνές ποινικό δικαστήριο. Πρόκειται για τροπολογίες για την παράγραφο 16 λοιπόν και οι τροπολογίες αυτές από την 109 στην 129 λέει η συγγήτρια είναι οι τροπολογίες αυτές που καλύπτουν αυτό το θέμα. Τώρα για τις τροπολογίες αυτές εγώ θα ήθελα να δώσω την πρέφουσα προσοχή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μέσα στα πλαίσια της αιτήσιας εκθεσής μας, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το κέριο, το κεντρικό θέμα στην αιτήσια εκθέση μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά όμως αξίζει την προσοχή μας και γι' αυτό εγώ θα καταθέσω ορισμένε προτάσεις συμβαστικού χαρακτήρα σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. <clears throat> Επίσης πρέπει να σας τονίσω ότι η περίοδος στην οποία καλύπτει η έκθεσή μας είναι από τα μέσα του 2008 μέχρι το τέλος του 2009. Επομένως και εγώ βασίζομαι στην κατανόησή σας. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε γεγονότα του 2010 εφόσον ενδιαφέρουν και την χρονική περίοδο που καλύπτω. Είναι δύσκολο όμως να αναφερθούμε σε θέμα του 2010 σε μια έκθεση η οποία καλύπτει το διάστημα μέχρι το 2009. Όσο σημαντικά είναι τα γεγονότα λοιπόν και οι συνδιασκέψεις που αναφέρονται, υπάρχουν και άλλα θέματα του 2010, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλω να τους αφαιρέσω το δικαίωμα να αναφερθούν σε αυτές τις <clears throat> παραβιάσεις, αλλά πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο, το χρονικό ορίζοντα της έκθεσης τελειώνει το 2009. Σας είπα λοιπόν ότι θα καταθέσω συμβασικές τροπολογίες για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσω να σας στείλω τις συμβαστικές τροπολογίες γιατί δεν έχουμε κάποια συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι αυτό μας δίνει τότε μία εβδομάδα μέχρι την ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θα μας δώσει αυτό τη δυνατότητα να επιληφθούμε των συμβαστικών τροπολογιών και να τις συζητήσουμε. Επίσης έχουμε τις τροπολογίες 142, 143 και 145 του κ. Χάουιτ, Ντόνσκης και άλλα που αφορούν την πυρικοποίηση τη ομοφιλοφιλία. Η διατύπωση τώρα αυτή τη τροπολογία είναι περίπου ταυτόσιμη. Επομένω, εγώ θα παρουσιάσω μια συμβαστική τροπολογία για τα θέματα αυτά. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, παράγραφος 21. Έχουμε τροπολογίες από την 161 ως την 168. αφορούν την ε, περιβόητη έκθεση Goldstone. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό που θα πω, αλλά εγώ πιστεύω το εξή ότι οι απόψει για την έκθεση Goldstone είναι ιδιαίτερα αποκλίνουσες μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και εγώ, σαν συμβαστική τροπολογία, θα ήθελα να προτείνω να μην κάνουμε καμία κρίση είτε θετική είτε αρνητική για την έκθεση Goldstone. Θα λάβω υπόψη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προσπαθήσω να απηχήσω και τις δικές σας προτάσεις όσο μπορώ καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπησέρθουμε σε μια αξιολόγηση της έκθεσης Goldstone. Αν δεν σας αρέσει μια τέτοια συμβαστική θέση, θα αναγκαστούμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε άλλες προτάσεις αργότερα για τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε 22 για τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μάλλον. Έχουμε περίπου 22 τροπολογίες. Θα διατυπώσω και εκεί κάποιες συμβαστικές τροπολογίες για τους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι διατυπώσεις σε όλες τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί είναι πολύ κοντά <clears throat> μεταξύ τους. Και επίσης θα προσπαθήσω να έχω θετικό πνεύμα και επικοδομητικό πνεύμα όταν αξιολογώ την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την προστασία των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και φυσικά θα προσπαθήσω να μην κάνω σχόλια και κριτικές που να μην έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα. Όταν αναφέρομαι σε συγκεκριμένε χώρε και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένε χώρε Ρωσία, Ιράν, Κίνα, Κούβα, θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν κατατεθεί κάποιες τροπολογίες για τις χώρες αυτές και εγώ θα προσπαθήσω να βρω μια συμβιβαστική πρόταση για τις χώρες αυτές, οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές μας συμφωνίες. Εδώ πρόκειται για το, την παράγραφο 60. Πολλές είναι τροπολογίες από τις 283 στις 285 καταρχήν θα προσπαθήσω να τις συγχωνεύσω σε μια συμβαστική τροπολογία. Υπάρχει και μια τροπολογία για την Κολομβία και μπορώ να φανταστώ ποια είναι η θέση της δικής μου πολιτικής ομάδος. Μόλον τούτο θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη την πρόταση αυτή που έχει γίνει για τροπολογία σε ό,τι αφορά την Κολομβία και να την ενσωματώσω στην ετήσια έκθεση. Θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης. Υπευλήθησαν και εδώ πολλές τροπολογίες. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να διατυπώσω μια συμβαστική πρόταση, αλλά θα πρέπει να καταγράψουμε τι χώρε οι οποίες, ε, ένα ερώτημα είναι αν πρέπει να καταγράψουμε όλε τι χώρε οι οποίε παραβιάζουν την ελευθερία θρησκείας. Επίση για την παράγραφο 73, οι τροπολογίε που αναφέρονται εκεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατία και το άρθρο, η παράγραφο μάλλον 74 είναι πολύ σημαντική γιατί αναφέρει τον όρμον του Ουαντάναμο, το κέντρο κράτησης, υπάρχει η τροπολογία του κ. Προβέρα όπου προτείνεται να βάλουμε και ένα νέο στοιχείο ε, στο, στην έκθεσή μας σε σχέση με τους σεξουαλικούς ακροτηριασμούς. Εγώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα χωριστό τμήμα στην ετήσια έκθεση για το θέμα αυτό. Σίγουρα όχι 7 παραγράφους για αυτό το θέμα. Οι τροπολογίες από το 2.01 ως το 2.07 καλύπτουν το θέμα αυτό και θα προσπαθήσω να τις λάβω όλες αυτές υπόψη. Τροπολογία 2.09 για την Νότια Αμερική αφορά τους φόνους ε, τρανσεξουαλικών ατόμων στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αμερική, συγγνώμη. Για τα φιλομεταβατικά αυτά άτομα νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και ίσως οι συνάδελφοι μπορούν να εκφράσουν καλύτερα τις απόψεις τους σήμερα για το θέμα αυτό εφόσον το επιθυμούν. και να εκφράσουν την άποψή τους για τις συγκεκριμένες χώρες οι οποίες αναφέρουν. Αυτά λοιπόν τα κύρια θέματα στα οποία εγώ ήθελα να εστιάσω στη σημερινή συζήτηση. Δεν ξέρω αν δέχεστε την προσέγγιση μου. Κύρια θέματα είναι διαθέσει ποινικό δικαστήριο, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένες μέρες περιπτώσεις σε διάφορες χώρες, Ρωσία, Ιράν, Κίνα και Κούβα ελευθερία θρησκευτικής ε, έκφρασης και άσκησης, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Αυτά τα κύρια θέματα που θέλω να αναφέρω. Η πρόεδρο έχει αναφέρει το χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα μα δίνει αρκετό χρόνο για συζήτηση μέσα στι πολιτικέ μα ομάδε. Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια να συναντήσω του κοιόδη συγγητέ από άλλε πολιτικέ ομάδε και να μπορέσω να συζητήσω μαζί του συμβαστικού χαρακτήρα τροπολογία. Πολύ καλά μα τα παρουσιάσετε. Απαντώντα για όλε τι τροπολογίε που κατατέθηκαν από ομάδε και συναδέλφου και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Ε, Mr. Mr και οποιονδήποτε άλλο, την κυρία Γέγκε, να λάβουν το λόγο. Κύριε Ντόντσκι πρώτος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την θαυμάσια παρουσίαση της εργασίας της ε, τη δουλειά που έκανα για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Εγώ έχω καταθέσει αρκετέ τροπολογίε που τονίζουν ορισμένα μηνύματα τη έκθεση. Παρόλο που είναι πάρα πολύ καλή έκθεση, νομίζω ότι έπρεπε να διευκρινίσουμε ε, τους χρήση κάποιων όρων. Να καλούμε το, το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων, των Ηνωμένων Εθνών να λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να καλούμε τα κράτη-μέλη και την ύπατη εκπρόσωπο να λειτουργεί με τρόπο που να καταστήσει τις ε, ενέργειες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιο, αποτελεσματική, πιο αποτελεσματικές και επίσης αναφερόμαστε στη, στη συνόδους των Ηνωμένων Εθνών και στις προτεραιότητες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. με τροπολογίες που υπογραμμίζουν τη σημασία, το ρόλο των ΜΚΟ για την ανάπτυξη και την προώθηση δημοκρατικών κοινωνιών και την προώθηση της ανεκτικότητας και της, του αμοιβαίου σεβασμού. Επίσης υπάρχουν ε, απειλές στην ελευθερία της επιστήμης επιστήμης, της συνείδησης και της γνώσης, της γενετήσου προσανατολισμού και επίσης και μια, ένα άλλο σημαντικό δικαίωμα που είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν όλα αυτά. Η αποδυνάμωση ειδικότερα των ευρωπαϊκών πολιτικών σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την κατάσταση στο Ιράν. Υποστηρίζοντα αυτέ τι τροπολογίε, νομίζω ότι θα κάνουμε μια ήδη πάρα πολύ καλή έκθεση, ακόμα πιο καλή και θα μεταφέρει ένα πιο ισχυρό, ισχυρό μήνυμα ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά έχω να προτείνω και ακόμα μια φορά συγχαίρω για το έργο τη την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κύριου Χάουιτ που δεν μπόρεσε να είναι παρόν, αλλά μπορώ να μεταφέρω τις απόψεις του μετά από αυτά που συζητήσαμε στην ομάδα μας. Φυσικά έχουμε μια θετική γνώμη για το σχέδιο έκθεσης και συγχαίρουμε την εισηγητρία. Πιστεύουμε ότι η προσπάθειά της εντάσσεται σε ένα σωστό πλαίσιο, αλλά όμως πρέπει να διευκρινίσω τη θέση μου. Σε ό,τι αφορά κάποιες προτεραιότητες ε, που πρέπει να αντανακλώνται. Καταρχάς, σε πολλά τμήματα του κόσμου υπάρχει πολύ άσχημη κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ορισμένε περιπτώσεις βελτιώνεται η κατάσταση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις προσπάθειες και θα πρέπει να το καταστήσουμε προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καταρχάς μέσω της ε, οριστικής κατάργησης θανατική ποινή. Το τελικό κείμενο μέσω των τροπολογιών θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτή. Καθώς και η υπεράσπιση των, των των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίσης μεγάλη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια δεύτερη ιδέα που θα πρέπει να απηχείτε στο τελικό κείμενο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια, μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δυστυχώς κάτι που, πρέπει να, κάτι που συνδέεται με αυτό. Ε, μεγαλύτερη συνέπεια σε ηθικό επίπεδο στον τρόπο που αντιδρούν, στον τρόπο που δρούν και αντιδρούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κατανέμουν μεταξύ τους τους ρόλους. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης, να δούμε τι γίνεται, όχι μόνο οικονομικός ρεαλισμός, θα πρέπει να υψώνουν και τη φωνή τους ε, όταν υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνέπεια λοιπόν τη δράση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλη ηθική ας πούμε και εδώ και άλλη εκεί. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένες χώρες με πολύ ξεκάθαρο τρόπο του κόσμου. Βεβαίω το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει που μπορούμε να καταγγείλουμε ή που πρέπει να καταγγείλουμε και επομένω θα πρέπει να ιεραρχήσουμε λίγο τι προτεραιότητέ μα. Η... Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στι πιο σοβαρέ περιπτώσει, τι πιο κρυφέ περιπτώσει και εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη αδυναμία. Και πολύ περισσότερα θύματα ή πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Και εκεί που υπάρχει δυνατότητα να επηρεάσουμε τα γεγονότα βέβαια. Αυτή είναι η θέση της ομάδας μας. Επίσης, κάτι άλλο. Θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι μπορεί να επηρεάσει πιο πολύ η έκθεσή μας τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Όμπιλς. Μιλάτε από την εμπειρία ε, του εισηγητή της προηγούμενης ετήσιας έκθεσης και όλοι συμφωνούμε με την εκκλησία σας για μια ισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και συγχαίρω την εισηγήτρια που την ετοίμασε με πολύ ε, ικανοποιητικό τρόπο και έτσι αποτελεί μια βάση για περαιτέρω συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω από 400 τροπολογίες πρέπει να το θεωρήσει ένα κομπλιμέντο η κυρία Ντρίκενε και ως θετική ανταπόκριση στην έκθεσή της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να παρουσιάσει μια ισχυρή έκθεση η οποία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την πιο αποτελεσματική πρόθεση αυτού του σημαντικού θέματος και θα ήθελα να κάνω και μερικές ακόμα παρατηρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο για τον, σε προγράμματα εκδημοκρατισμού και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα ωστόσο αυτών των προγραμμάτων δεν ήταν πάντοτε απόλυτα σαφή και ξεκάθαρα. Οι προσπάθειες πρέπει ωστόσο να συνεχιστούν. Η υποστήριξη του, τις διαδικασίε του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να συνεχιστούν παρόλο που έχουν διαταραχθεί οι ισορροπίε δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα. Μέχρι στιγμή, υπάρχουν ε, ε, δεσμεύσεις στα λόγια μόνο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μεταφράζονται σε πρακτικά αποτελέσματα και αυτό που λείπει είναι η παρακολούθηση αυτών των δράσεων. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδοντας στη, πιο δυναμική παρουσία και παρέμβαση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ενσωματώνονται στις δομές της υπηρεσίας αυτής και να αποτελέσουν μέρος των δραστηριοτήτων της. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ε, συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους τομείς εξωτερικής δράσης. Ανάπτυξη πολιτικής, ε, άμυνα, ε, εμπόριο κλπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει προβλήματα ε, συμμετοχής στις πληροφορίες και ενημέρωση για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σε άλλα θεσμικά όργανα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά πρέπει να επιμείνει για μεγαλύτερη διαφάνεια και πλήρη πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία και σε όλα αυτές τις αξιολογίες και τα έγγραφα που υπάρχουν σε άλλα θεσμικά όργανα. Διάλογο με τρίτες χώρες. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί το διάλογο και τις διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες. Ωστόσο πιστεύω ότι αυτός ο διάλογο και οι διαβουλεύσεις πρέπει να καταστούν πιο αποτελεσματικοί, να γίνεται σαστή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών των ε, επαφών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξακολουθεί να παρακολουθεί μη, ε, χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ισχύει για ευρωπαϊκές χώρες ειδικότερα που προσβλέπουν στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν συνεπείς στρατηγικές οι οποίες θα προβάλλουν την ανάγκη για τον εκδημοκρατισμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος θέλω να πω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση που μας παρουσίασε η συγγήτρια για το πώς θα αντιμετωπίσει ε, όλες αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτά που άκουσα από τους σκιώδεις εισηγητές και την αντικατάστασή τους ήταν θαυμάσιες δηλώσεις. Και θα μιλήσω την Πέμπτη στους 28 ακολούθους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης για να συζητήσουμε την αναθεώρηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά που άκουσα με έχουν ε, ευχαριστήσει πάρα πολύ και θα μεταφέρω το μήνυμα και στις, στα άλλα θεσμικά όργανα. Η κυρία Γέγλε και η κυρία Γκάλ επόμενες ομιλήτριες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία εισηγήτρια. Νομίζω ότι έχετε ήδη συντάξει μια πολύ καλή έκθεση καταρχήν και δεύτερον έχετε με όλες αυτές τις πολύ καλές τροπολογίες μια πολύ καλή ευκαιρία να προχωρήσετε, να δημιουργήσετε συμβαστικές τροπολογίες επί τη βάση της οποίας θα βελτιωθεί και η έκθεση αυτή πολλές τροπολογίες είναι απλώς διατύπωσης και μόνο. Φραστική δηλαδή τροπο, τροποποίηση, όπου ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και περισσότερο στο θέμα της σωστής μετάφρασης αυτών των διατυπώσεων. Να υπάρξει απαραίτητη μέρημνα ώστε να εκφραστούν σωστά στις αντίστοιχες γλώσσες. Και εσείς ήδη αναφερθήκατε στο θέμα αυτό της θρησκευτική ελευθερίας και της ελευθερίας έκφρασης. Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό και εγώ και να τονίσω τη σημασία του διαλόγου με τρίτες χώρες. Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση, την ακρόαση μάλλον εδώ χθες, και αυτοί οι οποίοι όπως εγώ είναι εδώ και χρόνια στην αντιπροσωπεία για την Κεντρική Ασία και γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση εκεί ή αν κάποιος ασχολείται με τα θέματα της Τουρκίας και είδε όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα έχουμε τονίσει στο παρελθόν και έχουμε κάνει αιτήματα σχετικά και δεν έχουν προχωρήσει κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν να μην σταματήσουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Ένα επίσης επιχείρημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό έχει να κάνει και με την ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία Δράσης. Και επίσης έχει να κάνει και με εμπορικές ή ακόμα και αγροτικές συμφωνίες. Εμείς κάνουμε λοιπόν πάρα πολλές συμφωνίες με τρίτες χώρες και θα πρέπει από τη δική μας πλευρά να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση αυτών των ε, συμφωνιών. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη επιρροή στη σύναψη αυτών των συμφωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορούμε να έχουμε γέρο τι πληροφορίε και να μπορέσουμε να παίξουμε κάποιο ρόλο στο περιεχόμενο αυτών των συνθηκών. Με την ανάγνωση τη έκθεση τη κυρία Ανδρίκαινα γίνεται αυτό πάρα πολύ σαφέ. Για μένα λοιπόν οι συμφωνίε ε, εταιρικού χαρακτήρα με χώρε τη Κεντρική Ασία ή με χώρε τη ε, Λατινική Αμερική είναι ακριβώς τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση γιατί θα μας δώσουν ενδεχομένω τη δυνατότητα να έχουμε κάποια επιρροή για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι άμεσα συνδεόμενο με την έκθεση της κυρίας Αντρίγκεν, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Στην περίπτωση του Καζακστάν, ας πούμε, είδαμε χθε ότι έχουν ληφθεί ήδη κάποιες νομοθετικές μέρημνες και πρόνοιες, αλλά στη συνέχεια στο επίπεδο της εφαρμογής δεν πραγματοποιούνται αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί στο χαρτί. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες αυτών των συμφωνιών <clears throat> για να πιέσουμε τους ε, συνομιλητές μας να <clears throat> εφαρμόσουν και στην πράξη όλες αυτές τις ε, συμφωνίες οι οποίες έχουν ε, διατυπωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γέγκλα. Νομίζω ότι θίξατε ένα σημαντικό σημείο τη στρατηγικής της υποεπιτροπής μας όταν τονίζεται την ανάγκη να είμαστε πιο πολύ εμπλεκόμενοι στη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνουμε και αυτά τα στοιχεία υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και προς την κατεύθυνση ορισμένων πιλωτικών σχεδίων και νομίζω ότι η άσκηση επιχάρτου ουσιαστικά που θα έχουμε στην περίπτωση της συμφωνίας εταιρικού χαρακτήρα με το Τουρκμενιστάν θα είναι και μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε πλήρως την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν περνάμε σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκμενιστάν. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αν αυτή η συνεργασία θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ε, πίεση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αν αυτά είναι απλώς ευσεβείς πόθη. Σας ευχαριστώ κυρία ε, Γέκλ και το λόγο στην κυρία Γκάλ. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την εισηγήτρια λέγοντας ότι είναι θαυμάσια η έκθεσή της. Οι πολλές τροπολογίες οφείλονται στη σημασία του θέματος και στη σημασία του μηνύματος που θέλουμε να μεταφέρουμε. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά τη διατύπωσή της, διότι πρέπει να μεταφέρει το σωστό μήνυμα. Έχουμε όχι μόνο υποχρέωση, αλλά και ευθύνη αναλάβει ετοιμάζοντας αυτή την έκθεση. και πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα ώστε τελικά να έχουμε μια εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριε Βεζιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να τη ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συμμετέχω στην τελευταία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Οι βοηθοί μου ωστόσο με ενημέρωσαν πλήρω για αυτά που ελέγχθησαν εκεί. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι για μένα υπάρχει μόνο μία προσέγγιση, μία αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι οικουμενικά, πρέπει να υπάρχουν παντού τα ίδια για όλους και αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερες υποχρεώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πω με κάπως προκλητικό τρόπο, η οποία μιλάει συχνά, αναφέρεται συχνά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μένει στα λόγια. Ενώ γιατί αν θέλουμε να προασπίσουμε και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό σημαίνει υποχρεώσεις που καλείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις με όλες τις τρίτες χώρες. Αυτό ελέγχθη ήδη, αλλά ξέρουμε ότι ορισμένα κράτη τα ε, περισσότερο σε ό,τι αφορά κάποιες τρίτες χώρες σε σχέση με άλλες. Δεν θα επανέλθω στο θέμα του βραβείου Ζαχάροφ, αλλά θα μιλήσω περισσότερο για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αφρικανικές χώρες. Με τις αφρικανικές χώρες πιστεύω ότι ε, έχουμε, πρέπει να αναλάβουμε ειδικέ υποχρεώσεις πολλές χώρες Αφρικής είναι δικτατορίες. Οι δικτατορίες αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν με την ε, υποστήριξη μεγαλύτερη μικρότερη ορισμένων κρατών μελών και με τη σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η σιωπή είναι βαριά. Είναι βαριά για τους υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αγωνιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι αγωνίζονται με εκείνο τη ζωή του, καθημερινά σε ορισμένε από τι χώρε αυτές. Και θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή τη σιωπή απέναντι σε αυτές τις χώρες. Οι σχέσεις που διατηρούμε με χώρες όπως η Λιβύη, την Ισία, είναι σε, από πολλές απόψεις μη παραδεκτές. Γι' αυτό, γι' αυτό και πάλι προκλητικά ε, έχουν συνηθίσει πια αυτοί που με γνωρίζουν καλύτερα. Δεν είναι μόνο οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι μουσουλμανικές χώρες. Παντού, παντού στον κόσμο πρέπει να υπερασπίζονται με τα ίδια ιδανικά, με βάση τα ίδια ιδανικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η οικουμενική αντίληψη για τα ανθρωπ τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά τόσο τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα όσο και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Και αυτό είναι και το νόημα κάποιων τροπολογιών που κατέθεσε. Αυτό σημαίνει η οικουμενική διάσταση. Το, το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεν είναι δυνατόν να τα διαχωρίσουμε τα δύο. Πολλές φορές προβάλλονται σε βάρο των ελευθεριών τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό το βλέπουμε σε πολλέ χώρε. Αυτές οι αξίες είναι εξίσου θεμελιώδεις όσο τα αισθητικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Τέλος, τελευταίο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, πάντα για να προβάλλω τις θέσεις μου. Η ελευθερία συνείδησης είναι, σημαίνει ελευθερία θρησκείας αλλά και ελευθερία του να πιστεύει να μην πιστεύει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να αποδώσουμε την ίδια σημασία σε εκείνους που απειλούνται επειδή δεν πιστεύουν. Η ελευθερία συνείδησης είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία του να πιστεύει κανείς ή να μην πιστεύει, του να επιλέγει μια θρησκεία, να, τη δυνατότητα να ασκεί αυτή τη θρησκεία. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συνόλου και με από αυτή την άποψη η έκθεση ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, οπωσδήποτε ε, επιδέχεται κάποιες βελτιώσεις, αλλά αν κάνουμε τις αναγκαίες προσπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ομοφωνία, σε σύμπτωση απόψεων, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο το μήνυμά μας, το μήνυμά μας θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό σημείο και ελπίζω να το συμμεριζόμαστε όλοι. Ε, ελπίζω να δείχνουμε ότι πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αυτό ε, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι την προσοχή μας την, την έχει όλος ο πλανήτης ε, ίσως βεβαίως ε, θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην Αφρική και να δουλέψουμε με την Επιτροπή Ανάπτυξης για να εξασφαλίσουμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Υποσαχάριο Αφρική αλλά και στην Βόρεια Αφρική. Τώρα, ως και όδηση συγγήτρια της ομάδας μου θα πω και εγώ δύο λόγια. Είμαι ικανοποιημένη που η συγγήτρια έδωσε έμφαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ίσως θα μπορούσε να απλουστεύσει τις ε, τροπολογίες, ε, ούτως ώστε να ενταχθούν στο στυλ και στο ύφος της έκθεσης. Δεύτερη παρατήρηση. Εκεί που αναφέρεται την έκθεση Goldstone και το θέμα της Κολομβίας που διαιρεί το Κοινοβούλιο, ελπίζω εμείς εδώ στην Υποεπιτροπή να δημιουργήσουμε μια στεναρή βάση, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις ε, πολιτικές διαφωνίες, τις κομματικές διαφωνίες και να εξετάσουμε το θέμα μόνο από σκοπιά ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτω ώστε να γίνουμε το βάθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είμαστε εμεί η καρδιά τη ε, πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Ε, ίδια κριτήρια σε ίδιε καταστάσει σε διάφορα μέρη του κόσμου. αυτή είναι, θα πρέπει να είναι η προσέγγιση μα. Αυτά που έχει ήδη πει το Κοινοβούλιο για την έκθεση Goldstone μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη μας. Η συγγήτρια θα αποφασίσει τι θα γίνει εν τέλει όμως. Ε, αυτά είχα να σας πω. Εσείς θα δείτε τώρα τι θα κάνετε με όλα αυτά τα σχόλια που ακούσατε. Α, είχα προσκαλέσει και την Κομισιόν να συμμετάσχει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Ενέ και για, να την συγχαρώ και για τον σημαντικό αριθμό των τροπολογιών. Από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, κάτι που δείχνει τον κεντρικό ρόλο και εκ των του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεισφορά του στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο. Θέλω απλώς να τονίσω ότι είμαστε ικανοποιημένοι για την εμβέλεια, την πολύ ευρεία της έκθεσης. Πολλά θέματα αναφέρονται στην έκθεση είναι ε, και στις πολυάριθμες τροπολογίες. Καταφέρνετε να καλύψετε το σύνολο του φάσματος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη και τα πιο πρόσφατα γεγονόματα ε, επί των οποίων δρούμε τώρα, παραδείγματος χάρη την ελευθερία της θρησκείας και, των πεπιθήσεων, σκεπτικών πεπιθήσεων. Όλα, παραπέμπω σε όλα αυτά που είπε η κυρία Βεωσία πριν από λίγο. Και η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ομοφιλοφίλους άνδρες και γυναίκες και τους φιλομεταβατικούς. Και εκεί επίσης εστιάζουμε τη δράση μας. Επίσης είμαι ικανοποιημένο για την προσοχή που δίνει η κυρία Αντρική Ενέ στην αποτελεσματικότητα της κοινή δράση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη και στα διάφορα βήματα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα εκεί τεκτενόμενα. Υπάρχει μια έκθεση παρακολούθησης για τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό και χαιρόμαστε που αναφέρεται την έκθεση Goldstone επίσης και οι υπόλοιποι ομιλητές την ανέφεραν και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ξεπέρασε τις εσωτερικές διαιρέσεις της για να αντιδράσει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα όσα αναφέρει η έκθεση Goldstone για το θέμα του στολίσκου και χαιρόμαστε που στην ε, Σύνοδο του Σεπτεμβρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε κοινή θέση, αποχή ήταν η θέση της, αλλά η θέση αυτή απηχεί μια ουσιαστική συμφωνία ε, και εξήγησε αυτή τη θέση με επεξήγηση, ε, με επεξήγηση ψήφου το Σεπτέμβριο στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκθεση Γκολστόν και για τον Στολίσκο. Επίσης, πέρα από την ε, αντίδραση από πλευράς μας στα στοιχεία της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη σε εσάς κύριε Αντρικίενε, αγγίζει τα ουσιαστικά θέματα της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, θυμάστε στις 16 Ιουνίου, κυρία Άστον, ε, έκανε μια έκκληση, μια αναγγελία μάλλον, ότι ξεκινάει μια διαδικασία διαβούλευσης, ούτως ώστε ε, να μεταρρυθμίσει την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης, ε, όπως είπε η κυρία Χαουτέλα, και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι κυρία είναι φαίνεται να είσαστε σε θέση να δημιουργήσετε ένα σημείο σύγκλησης ε, μεταξύ όλων αυτών των παρατηρήσεων που έχουν ακουστεί. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. <coughs> Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Αντρικίνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους από εσάς για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση αυτή και για την έκφραση ιδεών και σχολείων. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το εγχείρημα επί του οποίου εργαζόμαστε όλοι φυσικά δεν είναι απόλυτα τέλειο. Ελπίζω ότι πριν από τις 9 Νοεμβρίου που θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε ορισμένες συμβαστικές λύσεις και κυρίως με ενδιαφέρει η ανάδυση συμβαστικών λύσεων για τα πιο ευαίσθητα θέματα, γιατί έτσι μονάχα θα αποκτήσει προσθέμενη αξία η έκθεσή μας. Μου άρεσε η ιδέα που εξέφρασε η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Είπε ότι δεν είναι μονάχα μια ευκαιρία, αλλά και μια ευθύνη μας αυτή η έκθεση και κατανοώ απόλυτα ότι όλα αυτά τα οποία λέμε στην έκθεση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλα θέματα, για τα οριζόντια πρόβληματα, θα δώσουν ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς το σύνολο κόσμο για την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα τόσο σημαντικά αυτά θέματα. Θέλω επίσης να, εκφράσω και τις ευχαριστίες μου σε, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα άτομα και τους φορείς που έχουν έρθει σε επαφή με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της σύνταξης αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσά μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτές τις κοινέ λύσεις. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολλές φορές ακολουθούν πολύ αυστηρές πολιτικές θέσεις, κομματικές θέσεις, αλλά είναι οι αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας βοηθούν περισσότερο να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις. Οι σας λαμβάνονται ιδιαίτερα σοβαρά από εμά. Αυτό είναι και ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε κατά πόσο είναι σωστέ οι δικέ μα πολιτικέ θέσει ή όχι. Για κάποιε συγκεκριμένα τώρα ερωτήματα. Συμφωνώ γι' αυτό που είπατε ότι ή όχι. Για κάποια συγκεκριμένα τώρα ερωτήματα. Κύριε Οβιόλς, συμφωνώ για, ε, αυτό που είπατε ότι η κατάργηση της θανατικής ποινή είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας και εγώ δίνω μεγάλη έμφαση στο θέμα αυτό στην ε, ετήσια έκθεση. Επίσης για τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρομαι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανάγκη να υπάρξει συνοχή και αποτελεσματικότητα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι κομβική σημασία γιατί αν κάνουμε προτάσεις οι οποίες παραμείνουν στο χαρτί και δεν εφαρμοστούν ποτέ, όλα αυτά είναι ματαιότητες. Κύριε Ντόνσκης, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα καλά σας λόγια. Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά για μένα. Δεν αμφιβάλλω <clears throat> ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινέ συμβαστικέ λύσεις και εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα για τις προτάσεις που έχετε διατυπώσει, τις οποίες νομίζω μπορώ να αποδεχθώ αυτή την ίδια στιγμή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το ρόλο της υπά του εκπροσώπου και οι δύο αυτοί φορείς, οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Και τρέφω την ελπίδα ότι θα δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στα θέματα αυτά στην ετήσια Κυρία Γέγκλα αναφερθήκατε στις συμφωνίες εταιρικού χαρακτήρα και τις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχουν. Η εφαρμογή όλων αυτών των ρητρών που περιέχονται σε τέτοιες συμφωνίες πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντική και συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να επανέρχομεθα συνέχεια στα θέματα αυτά στις ετήσιες μας εκθέσεις. Ευχαριστώ και τον κύριο Κούκκαν για τα σχόλιά του. Και αυτά μπορώ να πω για την έκθεση αυτή και προσβλέπω σε μια συνεργασία μαζί σας επικοδομητική για τις συμβαστικές λύσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρος, κυρία Χάουταλ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για σε αυτή τη συζήτηση η οποία καταδεικνύει και ποια είναι η στατηγική μας για τα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων που όπως είπε και η κυρία Βεζιά θέλουμε να την ε, κάνουμε γνωστή όχι μόνο κύκλο ανθρώπων και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και τώρα θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι υπήρξαν κάποιες κάπως ανησυχητικές ειδήσει ή φήμες από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι δηλαδή <clears throat> οι αποφάσεις για τις δομές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει διεκδικήσει το Κοινοβούλιο επιμόνως, προς το παρόν αυτές οι δομές δεν φαίνεται να έχουν ένα προφανή χαρακτήρα. Με την άδειά σας λοιπόν θα στείλω μια επιστολή στην ύπατη εκπρόσωπο υπενθυμίζων εις αυτήν τι ακριβώς έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο από αυτήν και τον θεσμό τον οποίων επενδύεται. Ίσως θα είναι δύσκολο λοιπόν εκ των υστέρων να επηρεάσουμε τις δομές αυτές αν δεν δράσουμε τώρα. Αύριο ίσως είναι πολύ αργά, πρέπει να το κάνουμε σήμερα αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει να δώσει κάποια ε, σχόλια ή αν έχει κάποια αντίρρηση στο να γράψω εγώ μια επιστολή, αλλιώς θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε με το διευρυμένο προεδρείο σε μια ώρα ίσως. Κύριε Οβιόλ, θέλατε να πείτε κάτι. Όχι. Καλά. <clears throat> Εντάξει, οπότε μετά τις αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει θα, κάνω, θα συντάξω αυτή την επιστολή. Είμαστε σε προπορία χρόνου. Αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να συζητήσετε εδώ, έχουμε λίγα λεφτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω την ακρόαση για το Τουρκμενιστάν πριν από τις 10.30, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν μονάχα στις 10.30 και δεν έχουν έρθει και οι, οι ομιλητές μας ακόμα. Πάντα μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Κύριε Βερζιάτ. Θα έχουμε την ε, ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα στα πλαίσια του διευρυμένου προεδρίου. Ίσως να νομίζετε ότι έχω μονομανίες με, επειδή επανέρχομαι, αλλά η ακρόαση του Ευρωπαϊκού, Ευρωμεσογειακού μάλλον δικτύου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ακρόαση αυτή αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο, αν δεν απατώμε. θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε, Πρόεδρε, ότι θα την κάνουμε έγκαιρα, κυρία Πρόεδρε, αυτήν την ακρόαση. Κυρία Πρόεδρε, με ακούτε? Σε εσά απευθύνομαι, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα γίνει καθυστερημένα. Ξέρω ότι αναβλήθηκε αυτή η ακρόαση του Ευρωμεσογειακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν κατάλαβα καλά, όμως αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο αυτή η ακρόαση. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι πολύ αργά όταν γίνει αυτή η ακρόαση λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την, την, με την Τινησία. Μα ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα αυτό, καθώς και η κατάσταση στην Τινησία. Ο αριθμός των απεργών πείνας πολλαπλασιάζεται στην Τινησία. Θα ήθελα λοιπόν να δείξουμε την ίδια προσοχή σε όλους τους απεργούς πείνας. Uh, uh, η Τινησία, κυρία Βερζιά, λέει η Πρόεδρος, είναι σημαντική για την υποεπιτροπή μας. Σήμερα το πρωί είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων, ε, δηλαδή κάναμε ερωτήσεις και απαντήσεις ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το άρθρο 61α του, του ποινικού συγγνώμη, κώδικα, καθώς και για το πάγωμα κάποιας χρηματοδότησης ε, δυνάμει του μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όντω θα αναβλήθηκε αυτή η ακρόαση, αλλά βλέπετε ότι οι ατζέντε μας είναι πολύ γεμάτες. Πρέπει να ετοιμάσουμε και την αντιπροσωπεία που θα επισκεφτεί την Τινησία. Έχουμε πολλή δουλειά και ελπίζω ε, σε αυτή την προετοιμασία να συνεισφέρετε ενεργά. Να κάνουμε διάλειμμα. Um, uh, Uh, Ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Βερζιά για τη διαδικασία για το βραβείο Σαχάροφ. Νομίζω ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Ολομέλεια. Ο πρόεδρος ζήτησε νέες ιδέες για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε τη διαδικασία, ούτως ώστε να είναι αποδεχτή από όλους τους ευρωβουλευτές. Κυρία Βεργιά, κάνετε μια θαυμάσια πρόταση και ελπίζω η Υποεπιτροπή να συνεισφέρει στη συζήτηση για την μεταρρύθμιση της διαδικασίας για το βραβείο Ζαχάροφ. Κύριε Ομπιόλς, έχουμε λίγο χρόνο. Για τα τελευταία που είπαμε, για τη δυνατότητα να συνεισφέρει η υποεπιτροπή μας, ούτως ώστε να βρεθεί μια άλλη μέθοδος για το βραβείο Ζαχάροφ. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και μάλιστα είναι και επίγον. Έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο μέχρι τον, το επόμενο βραβείο. Έχουμε χρόνο να προβληματιστούμε και να πείσουμε μεν τους δε, ούτως ώστε να υπάρξει μια συνένεση. Αλλά νομίζω η σημερινή μέθοδος ε, επιτρέπει σε ορισμένα λόμπι να επιβληθούν ακόμα και στην πλειοψηφία. Έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και πολύ πρόσφατα. Αυτή είναι η σημερινή μέθοδος. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη για να κερδίσουμε την έγκλη που μας αξίζει κάτι τη χορήγηση του βραβείου Ζαχάροφ. Η υποψία και μόνο ότι γίνονται διολυστήσεις ή ότι Υπάρχουν και άλλα κίνητρα πέρα από τη διάθεση να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι στυλιτεύουν τη διαδικασία για το βραβείο. Καλό θα ήταν στην υποεπιτροπή μας λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένες διαδικαστικές ε, προτάσεις για να ξεπεράσουμε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο διευρυμένο Προεδρείο, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορούμε να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Ε, οι υπόλοιποι βλέπω ότι γνέφουν α, καταφατικά. Αυτό που θέλουμε είναι αξιοπρέπεια γύρω από την διαδικασία του βραβείου. Μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε την ακρόασή μας για το, το Τουρκμενιστάν. Ελπίζω να είναι εδώ όλοι οι ομιλητές. Βλέπω την ε, κυρία Χέιλ, βλέπω την ε, κυρία Μπέρκ, βλέπω την εισηγήτρια, βλέπω πολύ κόσμο. Προσπαθούμε να διορθώσουμε μια δυναμία να έχει ρωμανική διερμηνία η κυρία Νικολάη. Uh, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχουμε φτάσει στο θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης και έχω να σας κάνω μια πρόταση σχετικά με την διερμηνία στα Ρουμάνικα και από τα Ρουμάνικα. Uh, um, uh, η πρόταση είναι η εξής θα ακούσουμε τους εξωτερικούς ε, εμπειρογνώμονες και τους άλλους φορείς, τους άλλους οργανισμούς, ενώ ε, στο μεταξύ οργανώνουμε και την διερμηνία προς Ρουμάνικα, από Ρουμάνικα. Από Ρουμάνικα σε αυτή τη συνεδριάση, διότι η κυρία ε, Νικολάη πολύ δικαιολογημένα θέλει να μιλήσει στα Ρουμάνικα και θα το οργανώσουμε αυτό. Συμφωνείτε λοιπόν να αρχίσουμε τους άλλους ομιλητές. Αυτή η ακρόαση είναι αποτέλεσμα μια συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη σύνδεση, συμφων... Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκμενιστάν για την οποία θα ε, πάρει θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κυρία Νικολάη είναι η συγγήτρια για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία αποφάσισε ότι προτού ψηφιστεί το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η υποεπιτροπή θα μπορούσε να οργανώσει μία ακρόαση για τις προοπτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωσή του στο Τουρκμενιστάν και κατά πόσο θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την υπογραφή αυτή της συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία. Και αυτή πιστεύω ότι είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούμε από εδώ και πέρα στο Κοινοβούλιο για τι σημαντικέ διεθνεί συμφωνίε. Η Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία υπεγράφει το 2008 και βρίσκεται 98, συγγνώμη, 98 και βρίσκεται ακόμη υπό τη διαδικασία επικύρωση. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα, την, την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να εγκρίνει τον Ιούλιο του 2009 την ε, ενδιάμεση συμφωνία και η συμφωνία φτάνει στην τελική της φάση. Πρόσφατα ξεκίνησε η εφαρμογή της σε δύο, στις δύο ε, ξανατέθη το θέμα στις δύο χώρες, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν την έχουν ακόμα επικυρώσει και καλείται λοιπόν και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του, τη σύμφωνη γνώμη του. Η σύμφωνη γνώμη λοιπόν του Κοινοβουλίου απαιτείται. Και όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του στην ενδιάμεση εμπορική συμφωνία τον Απρίλιο του 2009, το Κοινοβούλιο είχε θέσει ορισμένους στοχοδείκτες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει πρώτον ανεφόρον απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, κατάργηση όλων των εμποδίων στο ελεύθερο εμπόδιο, ελεύθερη πρόσβαση σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα παρακολουθούν την κατάσταση, ε, βελτίωση των ε, πολιτικών ελευθεριών και για ΜΚΟ ειδικότερα, η δυνατότητα της κοινωνίας των πολιτών να αναπτύσσεται χωρίς κρατηρικές παρεμβάσεις ε, θρησκευτική ελευθερία και ανοιχτές και αδιάβλητες και ελεύθερες εκλογές. Το μήνυμα του Κοινοβουλίου ήταν απόλυτα σαφές αυτή η ενδιάμεση συμφωνία δεν θα ήταν μια επιταγή εν λευκό. Απαιτούσε τακτικές ε, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις και παρακολούθηση των θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν και αυτή η ακρόαση έχει σκοπό να ενημερώσει τα μέλη μας για το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα εν ώψη της ε, σύμφωνης γνώμης που θα δώσει για την ε, συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασίας στο Κοινοβούλιο. Μια προσωπική περίπτωση. Ο κύριος Φάρετ Μπατούλιν είναι ακτιβιστής υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποχρεούνται να κατοικεί εκτός του Τουρκμενιστάν για λόγους ασφάλειας, προσωπικής του ασφάλειας. Έχουμε λάβει πολύ σοβαρέ ε, σοβαρές πληροφορίες από διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ο κύριο του απειλείται σοβαρά. Σήμερα λοιπόν έστειλα μια επιστολή στον πρέσβη και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάγκη να μεριμνήσουν ο κύριος Φαρέτ Μπατούριν που κατοικεί εξ όσων γνωρίζω τώρα στην Αυστρία να μην απειλείται πλέον με κανένα τρόπο. Και ελπίζουμε ότι η περίπτωση αυτή θα δείξει ότι μπορούμε, μπορούμε κάτι να κάνουμε για να προστατεύσουμε έναν σημαντικό υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, έρχομαι στους ομιλητές. Έχουμε την κυρία Ζακλίν Χέιλ, την οποία ακούσαμε ήδη χθε όταν είχαμε την ακρόαση για το Καζακστάν, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής του Open Society Institute. Θα της δώσω λοιπόν το λόγο για 10 περίπου λεπτά και μετά τη χθεσινή εμπειρία πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα για μια ζωντανή συζήτηση αν δεν ξεπερνάτε, αν δεν ξεπερνάτε το χρόνο αγόρευσης που σας έχουμε δώσει με αποτέλεσμα τελικά να μην έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να λάβω τα Ελλάδα. σήμερα. Θα ξεκινήσω τα σχόλιά μου με δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν ότι το Τουρκμενιστάν είναι μια κακοδικούμενη αυταρχική χώρα και όχι ένας εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, ότι η συνεργασία με το Τουρκμενιστάν μπορεί να οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και να υποσκάψει και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλεξάνδρ Μουράτη Τσίεφ ήθελε να φύγει από το Τουρκμενιστάν να βρει εργασία γιατί δεν είχε το δικαίωμα να εργάζεται μέσα στην χώρα αυτή. Τον Ιούνιο του 2010 μετά από πολλέ προσπάθειες να πάρει την άδεια από τι υπηρεσίες μετανάστευσης του Τουρκμενιστάν αυτοκτόνησε. Απλώς δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Ήταν σε απόλυτο αδιέξοδο. Η κυβέρνηση είχε καταδιώξει την οικογένειά του προσπαθούσαν να πείσουν την μητέρα του που ήταν δημοσιογράφος να την διώξουν από τη θέση εργασίας. Αυτή η μορφή συλλογικής τιμωρίας που ασκείται στο Τουρκμενιστάν είναι πολύ χειρότερη και από άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Ο Μπατούλεν επίσης, του Μπατούλεν, είναι μία από τις ελάχιστες αξιόπιστες αντιφρονούντες απόψεις που εκφράζονται στο Τουρκμενιστάν και πηγή πληροφοριών για τον έξω κόσμο. Και τώρα οι αρχές προσπαθούν να τον κάνουν να σιωπήσει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Τουρκμενιστάν. Θέλω να χρησιμοποιήσω λοιπόν το σύντομο χρόνο μου να τονίσω ότι μια συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα με το Τουρκμενιστάν όχι μόνο θα υποσκάπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι και ένα στρατηγικό σφάλμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα τονίσω ότι δεν είναι πιστικά τα επιχειρήματα για μια εταιρική σχέση για να υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία με ένα τέτοιο εταίρο χωρί να θέσει ένα αμφιβόλο την αξιοπιστία τη και το κύρο τη. Θέλω επίση να διαφωνήσω με το επιχείρημα ότι με την εταιρική συμφωνία θα υπάρξει δυνατότητα να βελτιωθεί ο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο με το Τουρκμενιστάν. Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην συμφωνία λοιπόν κάνει απόλυτα παράλογο μια, το να έχουμε μια τέτοια άποψη. Δηλαδή να υπογράψουμε τη συμφωνία χωρίς να έχουμε καμία εγγύηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί και οι δύο πλευρές δεσμεύονται από αυτήν την συμφωνία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπάρχει και δυνατότητα αναστολή εάν δεν υπάρχει σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλά αν είχε κάποιο νόημα αυτή η συμφωνία, πριν στεγνώσει το μελάνι πάνω στην υπογραφή αυτή τη συμφωνία, θα έπρεπε να ανασταλεί αυτή η συμφωνία ήδη λόγω παραβιάσεω ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα προτού υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα και σταθμά που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006, 2008 και 2009 θα πρέπει να είναι το οδηγό νήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πρόωρο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει μια νέα νομική βάση μετά από την εμπορική συμφωνία που έχει ε, συναυθεί πέρσι και αυτό χωρίς καμία αξιολόγηση από την Κομισιόν. Σας υπενθυμίζω ότι η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία έχει μια ταυτόσημη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η συμφωνία αυτή που προτείνεται να συναυθεί που δεσμεύει συμβατικά το Τουρκμενιστάν για το σεβασμό των υποχρεώσεών του. Το 2009, για να μπορέσει να επιτύχει τη Συμφωνία του Κοινοβουλίου, η Κομισιόν ε, δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει βελτίωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν μέχρι την υπογραφή ε, της Συμφωνίας Εταιρικού Χαρακτήρα, καλύπτοντας και τα απαιτούμενα του Κοινοβουλίου. Προτού λοιπόν πιέσουμε για μια νέα εταιρική συμφωνία, θα πρέπει να καταδείξει η Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι το Τουρκμενιστάν πράγματι έχει κάνει κάποια πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτή και ότι φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει πίεση στην Ασκαμπάν. Σε πρακτικό επίπεδο, η Συμφωνία Συνεργασία και Εταιρικού Χαρακτήρα δεν είναι, ένα εργασίο, δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο θα οδηγήσει σε μεγάλα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει ήδη από το 2007 με το Τουρκουμενιστάν χωρίς εταιρική σχέση και συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δημιουργήσει προγράμματα δημιουργία ικανότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Σεπτέμβριο του 2010 με την UNDP, την Υπηρεσία Ανάπτυξη των Ηνωμένων ε, Εθνών και το Εργαλείο για τη Δημοκρατία, χωρί όμω μια τέτοια εμπορική συμφωνία. Ακόμα και η συνεργασία για την οποία μπορεί να ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συνεργασία έχει ήδη λάβει χώρα εκτό μια συμφωνία επί τη βάση ενό μνημονίου κατανόηση και αυτό ακολουθεί <clears throat> παρόμοιε συμφωνίε με άλλε χώρε τη περιοχή όπω το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Όλα αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται νέο νομικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω τεχνικών προγραμμάτων τεχνική αρρωγή. Κοντολογής η ικανότητά μας εργασίας στην χώρα αυτή δεν θα πρέπει να ατενιστεί ως μια δυνατότητα συστημικής προόδου και μια ευκαιρία για πρόοδο στη χώρα αυτή. Θέλω λοιπόν να τονίσω και το τρίτο σημείο το οποίο με ενδιαφέρει. Προβάλλεται το επιχείρημα ότι η Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικού Χαρακτήρα θα δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τουρκμενιστάν. Αυτό όμως το διαψεύδει η εμπειρία μας σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια συμφωνία αυτού του είδους με το Ουσμπεκιστάν για πολλά χρόνια και ακόμα δεν υπάρχει μια πλήρης αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα είναι πιο εύκολο να γίνει η πραγματικότητα στο Τουρκμενιστάν. Στο δε Τατζικιστάν από το 2003 υπάρχει υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να υπήρχε προηγουμένω συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικού χαρακτήρα. Επομένω, δεν είναι αυτό το κριτήριο το αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συμφωνία με τις χώρες αυτές, αλλά το πόσο το επιθυμούν οι ίδιες αυτές οι χώρες να έχουν καλύτερες επαφές. Αν θέλει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μεγαλύτερη παρουσία στο Τουρκμενιστάν, Τη στιγμή που οι ομάδε τη κοινωνία των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο Τουρκμενιστάν χωρί να υφίστανται απειλέ στη ζωή του, είναι πραγματικά ασαφέ ποιοι θα ήταν οι εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή και ποιε θα ήταν οι συνέπειε για την ασφάλεια και τη ζωή του και επίση και για το κύρο και την ακαιρεότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι έχουν πει οι εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν έχουν επίσημο χαρακτήρα, υπάρχει ήδη μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαίδευση ε, της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορίζονται από την ίδια την κυβέρνηση να εργάζονται όλοι αυτοί μονάχα με άτομα, κυρίως δημοσιογράφους, διαπιστευμένους στην κυβέρνηση. Επομένως όλη η διαδικασία στο Τουρκμενιστάν ελέγχεται από, τις, από την προεδρική εξουσία και είναι πολύ λίγα τα αυτά τα οποία μπορεί να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει αποτέλεσμα σε αυτό επίπεδο. Δυστυχώς είδαμε στο Τουρκμενιστάν ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε δράση της κοινωνίας των πολιτών αν η κυβέρνηση δεν επιτρέπει ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών και αν δεν τους επιτρέπει να ταξιδεύουν, να συνεταιρίζονται, να εκφράζονται τις απόψεις τους, να συναντούν συνομιλητές. Αν κάθε φορά ο κατάλογος των παρόντων και η ατζέντα καθορίζεται από την κυβέρνηση, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίζει ότι θα μπορέσει με τέτοιου είδους συζητήσεις και συναντήσεις να επηρεάσει τα πράγματα. Κοιτάξτε πώ είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί στο Τουρκμενιστάν, μάλλον οι εταιρείε τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Το Μάρτιο της, ε, του προηγούμενου έτου, ο επικεφαλή μια γαλλική κατασκευαστική εταιρεία πρόσφερε ένα στόλο αυτοκινήτων στον πρόεδρο του Τουρκμενιστάν για να μπορέσει να αποσπάσει μια συμφωνία για την εταιρεία του. Επίση, θέλω να αναφερθώ και στην εμπειρία των ιατρών χωρί σύνορα ήταν <clears throat> μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έφυγε από τη χώρα μετά από 10 χρόνια εργασίας γιατί ανημένα θα ήταν υποχρεωμένοι να παραβούν τις ίδιες τους τις αρχές. Τους ζητήσανε να είναι παρόντες και να παρακολουθούν ε, ενώ η υγειονομική ε, υπεύθυνοι της χώρας μαγείρευαν τις στατιστικές για τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές αρρώστιες. Αναγκαστήκαν τελικά να φύγουν από τη χώρα. Και αυτό μας φέρνει στο στρατηγικό θέμα των benchmarks, των, ε, της βαθμονόμησης και των κόκκινων γραμμών σε σχέση με τη στρατηγική μας. Χωρίς τέτοια ε, χωρίς τέτοιες κόκκινες γραμμές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό, πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρίνει τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρατήσει επαφές με τον Τουρκμενιστάν τα τελευταία χρόνια. Με, δια, με την διαμεσολάβηση του, μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Τουρκμενιστάν, με την παρουσία του Επιτρόπου Οτιγκέρ το, την άνοιξη του 2010. Όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς καμία συμφωνία συνεργασίας και, και ε, εταιρικού χαρακτήρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χαράξει καμία στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Τουρκμενιστάν και η τρέχουσα προτινόμενη συμφωνία δεν προτείνει κανένα τέτοιο πλαίσιο. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση που θέλουμε να έχουμε σε 5-10 χρόνια στο Τουρκμενιστάν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα ενισχύσει τι θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, θέλω να σχολιάσω γενικότερα την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσει όπω το Τουρκμενιστάν θα πρέπει να καταδείξουν τη θέλησή του να συνεργαστούν με την διεθνή κοινότητα μέσω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που θα βοηθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεργασία και σε άλλου τομεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να έχει και μια προοπτική που δεν περιορίζεται μονάχα σε μια κοντόφθαλμη στρατηγική που βασίζεται στις πηγές ενέργειας και τις αγοράς ενέργειας. Μια στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει το Τουρκμενιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί με ποιο τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους όπως τον Μοχάμετ Μουράτιεφ, τον Χατζίεφ και τον Τουχ Μπατούλιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη Jacqueline Χέιλ. Τώρα ακούσαμε από το Open Society Institute που έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά σε όλη αυτή την περιοχή. Υπάρχει πλέον διερμηνία προς και από Ρουμάνικα φαντάζομαι. Οπότε θέλει λοιπόν να πάρει το λόγο η συγγήτρια τώρα ή μετά την Επιτροπή τώρα. Πολύ ωραία. Και η πρότασή μου είναι να ακούσουμε μετά την εισηγήτρια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την Human Rights Watch και κατόπιν θα ακολουθεί η συζήτηση. Κυρία Νίκολάη, ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα, θα προτιμούσα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι το Τουρκμενιστάν δεν, στο, στο Τουρκμενιστάν δεν επικρατεί μια ιδανική κατάσταση και αυτό εξαρτάται από εμά. Εξαρτάται από εμά αν θέλουμε η χώρα αυτή να δώσει μια ευκαιρία στους πολίτες της να έχει πρόσβαση άμεση σε, στις άλλες, σε δημοκρατικές χώρες γιατί βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση σήμερα το Τουρκμενιστάν. Συνδέεται αυτό εν μέρη με την ιστορία του και θα προσπαθήσω να εξηγήσω, το εξηγήσω αυτό με την, σαν αποτέλεσμα της κομμουνιστικής ε, κληρονομιάς και λόγω της ε, έλλειψης πριν από τη δικτατορία ε, πολιτικής ε, κουλτούρας ε, σε αυτή τη χώρα όπου παραβιάζονται διαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο από τις αρχές αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες σε καθημερινή βάση. Το Τουρκμενιστάν είναι μια χώρα η οποία έχει μπει σε μια πορεία μεταρρύθμισης. Μια χώρα που έχει αντιληφθεί ότι πρέπει πλέον να σέβεται κάποιου δημοκρατικούς κανόνες σε διεθνές επίπεδο. Και δεν συμφωνώ με εκείνου που συγκρίνουν το Τουρκμενιστάν με τη Βόρεια Κορέα ή τη Βερμανία. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω κάνει έρευνες για το θέμα αυτό. Έχω μεταβεί στο Τουρκμενιστάν επίσης και έτσι έχω μια σαφή άμεση εικόνα του τι συμβαίνει και δεν μπορούμε ως εκ τούτου από ό,τι διαπιστώνω να συγκρίνουμε τη Βόρεια Κορέα παραδείγματο χάρη του Τουρκμενιστάν. Το, τη, η διακυβέρνησή τους την αφημιώνουν με μια δημοκρατική εντολή αλλά υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση για την περίοδο Ναζιόφ και η κυβέρνηση προσπαθεί να συνάψει μια δημοκρατική συμφωνία, ένα δημοκρατικό συμβούλιο με την κοινωνία προσπαθώντας να εξασφαλίσει για τους πολίτες ε, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και όλα αυτά σε ένα πιο σύνθετο πλαίσιο. Πολύ πρόσφατα το Τουρκμενιστάν υπέγραψε και επικύρωσε διεθνείς συμβάσεις, διεθνείς συμφωνίες αν κάποιος έχει την περιέργεια και θέλει να διαβάσει ένα σύνταγμα που μοιάζει πάρα πολύ με άλλα συντάγματα σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές του διατάξεις, αν έχει κάποιος αυτή την περιέργεια θα διαπιστώσει πώς έχουν τα πράγματα όπως και άλλες χώρες οι οποίες δήθεν σέβονται ε, τους δημοκρατικούς κανόνες διαπιστώνουμε υπάρχει τεράστια διαφορά αυτά, ε, ανάμεσα αυτά που αναφέρονται στο χαρτί και την πραγματικότητα. Εγώ ανήκω σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν και ξέρω ότι στη δική μου χώρα, αντιλαμβάνομαι ότι και στη δική μου χώρα για υποχωρούμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πολλών δημοκρατικών κανόνων και ανεχόμαστε ορισμένα πράγματα που δεν θα έπρεπε κανονικά να ανεχόμαστε. Για τις παραβιάσεις ωστόσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν αυτές πιστεύω ότι αφορούν το μη σεβασμό του κράτους δικαίου όχι με την έννοια που ε, δίνει σε αυτό το θέμα η ευρωπαϊκή παράδοση η ελευθερία ε, ε, κυκλοφορίας, η νομική προστασία σε περίπτωση δίκης, το δικαίωμα προσφυγής, η έφεση, άσκηση έφεση δεν τηρούν όλους τους κανόνες, αλλά γίνονται προσπάθειες προκειμένου να εγγυηθεί ο σεβασμός των ε, διαδικασιών, διαδικασιών της υπεράσπισης, ώστε να έχουν, μπορούν να, να, να έχουν μια δίκαιη δίκη οι κάτοικοι της χώρας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές ελευθερίες των πολιτών και αυτές παραβιάζονται και όλα αυτά συνδέονται με τη μακρά περίοδο δικτατορίας που επηρέασε, επηρέασε την ε, χώρα και τους κατοίκους της πριν και μετά την κομμουνιστική περίοδο. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να βοηθήσουμε το Τουρκμενιστάν να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις ε, αναμεταδόσεις των μέσων ενημέρωσης. Στο Τουρκμενιστάν παραβιάζεται λοιπόν η ελευθερία του τύπου, οι κάτοικοι δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τον τόπο κατοικίας τους, δεν τηρούν ορισμένα οικονομικά δικαιώματα επίσης. Υπάρχει λατρεία προσωπικότητας η οποία έχει μεταφερθεί από, προηγούμενη από το προηγούμενο στο σημερινό καθεστώς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κυβέρνησης του Τουρκμενιστάν ο πρόεδρος της χώρας ακολούθησε μια επαγγελματική δραστηριότητα διαφορετική από τους προκατόχους. Ήταν ιατρός, δεν ανήκει στην κομμουνιστική ελίτ όπως ο Νιαζόφ την εποχή του. Σήμερα μπορούμε νομίζω να πούμε το Τουρκμενιστάν προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτό το σκοτεινό του παρελθόν. Αυτό, προϋποθέτει, αυτό σημαίνει, συνεπάγεται πολλές δυσκολίες, διότι το σύστημα Νιαζόφ που ήταν ένα παρανοϊκό θα έλεγα σύστημα με φοβερές κυρώσεις σε τεράστια κλίμακα ήταν πάρα πολύ σκληρό για όλους στη χώρα. Ο ποινικό κώδικας, ο κώδικας ποινική διαδικασίας του κράτους τηρούν τους δημοκρατικούς κανόνες αλλά για κάποιους ανώτατους αξιωματούχους του, Αφγανιστα... του Τουρκμενιστάν η κατάσταση δεν είναι και τόσο ρόδινη. Οι συνάδελφοι της Human Rights Watch και του Open Society Institute αναφέρθηκαν ήδη σε αυτό και ασφαλώς θα μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατυπίστωσαν και ανακάλυψαν στο Τουρκμενιστάν. Πάντω το Τουρκμενιστάν ακολουθεί μια πορεία μεταβατική, μια πορεία μετα μεταρρύθμισης οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα ώστε να ακολουθήσει μια, μια νέα κατεύθυνση η χώρα σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, για την έκθεση που μου ανατέθηκε να ετοιμάσω, θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Τι καινούριο μπορεί να φέρει ε, μια τέτοια ε, έκθεση για να προσδιορίσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το Τουρκμενιστάν. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας μπορούμε να επιφέρουμε μια σειρά από καινοτομίες στον τρόπο που λειτουργούμε και ενεργούμε. Εγώ ζήτησα μια αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια της συμφωνίας. Ζήτησα το Κοινοβούλιο να εμπλακεί στην όλη αυτή διαδικασία και ζήτησα αυτή η αναθεώρηση να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στη συμφωνία σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταχρήσεις περιόρισε τη συμφωνία σε την ε, έκθεση σε ορισμένες σελίδες και ε, απίτησα να υπάρχει τερκής παρακολούθηση του εισπρόδου και επέμεινα στην ανάγκη να υποβάλλονται ε, συστάσεις στην κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν σχετικά με την στρατηγική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι αυτό θα υποστηριχθεί από όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι κατά πόσο ευθύνεται, πρέπει να θεωρήσουμε ότι ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι ο Τουρκμενιστάν δεν έχει τηρήσει, δεν έχει τηρήσει τις διατάξεις ε, των διαφόρων συμφωνιών. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ευθύνη ε, είναι κοινή και για τις δύο πλευρές. Γι' αυτό προτείνω και ένα μηχανισμό ταχείας αντίδρασης που θα χρησιμοποιηθεί αν διαπιστωθούν ε, παραβιάσεις των διατάξεων της συμφωνίας. Ένα άλλο θέμα που με απασχόλησε ήταν η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στο Τουρκμενιστάν. Αυτή είναι μια νέα διάταξη. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας όταν εργάζονται σε χώρες, σε περιοχές ευαίσθητες όπου υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι. Προσωπικά πιστεύω ότι οι προσπάθειες, όποιες και να είναι αυτές, για το Τουρκμενιστάν πρέπει να αφορούν κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να τιμωρήσουμε το του Τουρκμενιστάν επειδή είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς σπόρους. Δεν πρέπει να τιμωρούμε τους πολίτες του και να να τους, ε, χωρίς να τους επιτρέψουμε να ονειρεύονται μια καλύτερη και πιο αξιοπρεπή ζωή έστω και με τον κίνδυνο να φανούμε υποκριτές. Για το οικονομικό σκέλος πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε τη διαφάνεια. Αυτό κατά την άποψή μου είναι σημαντικό κριτήριο πρέπει να συζητούμε περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο υπογράφουν συμφωνίες τα κράτη-μέλη, κερδοφόρες συμφωνίες με τις χώρες της περιοχής. Ο μηχανισμός ε, ε, ε, Extractive Industries Mechanism είναι ένας μηχανισμός στον οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς μια συμφωνία τέτοιου είδους θα μπορούσαμε να εξακολουθούμε να περιμένουμε, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αντίδραση ή να έχουμε μια μόνο περιορισμένη αντίδραση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση και να αλλάξουμε και την προσέγγιση μας για τέτοιου είδους συμφωνίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπωσδήποτε πρέπει να σέβεται αφενός τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά να ενεργήσει, να αναλάβει δράση, πιο ενεργό δράση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποιες περιοχές και εγώ αισθάνομαι κάπως ένοχη ως Ευρωβουλευτής. Αισθάνομαι ένοχη για το γεγονός ότι δεν έχω καταφέρει να αναπτύξω σημαντικότερη δράση για μια υπόθεση τόσο σημαντική όσο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί ασφάλειας που ε, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν μια τέτοια συμφωνία διότι ε, αλλιώς με άλλο τρόπο δεν θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε την, να το σεβασμό των ανθρωπίνων Πρέπει να σας διακόψω γιατί πρέπει να εξασφαλίσω και χρόνο για τους υπόλοιπους ομιλητές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είχε παρακολουθήσει ε, εκ του σύνεγγυς ε, τι συνέβη με τα benchmarks ε, μεταξύ των ετών 2006, 2008 και 2009. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να μας πει, μετά από το Human Rights Watch. Επίσης, ο Ήπατος Επίτροπος εκπροσωπείται εδώ από το ΟΗΕ. Ο κύριος Άρβινσον, και η κυρία, συγγνώμη, Άρβινσον. Ε, ούτως ή άλλως εκπροσωπεί εδώ τον ΟΗΕ και έχουμε στενές επαφές με το γραφείο τους στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Γκούνα ε, Βίγκαν είναι ο Διευθυντής ε, Ανατολικής Ευρώπης, ε, Νότιου Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Χάουτελα που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα του Τουρκμενιστάν ε, εν ώψη τη επικύρωση τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία ε, με το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστώ, κύριε Νικολάη, για την προσπάθειά σα για να συντάξετε αυτό το σχέδιο ψηφίσματο. Θα ήθελα πολύ σύντομα να υπενθυμίσω ότι εδώ μιλάμε, όπω σωστά είπε και η Πρόεδρο, όχι για την υπογραφή μια συμφωνία, αλλά όπω είπε και η κυρία ε, Χέιλ, για την οριστικοποίηση μιας μακράς διαδικασίας επικύρωσης. Η υπογραφή έχει γίνει το Μάρτιο του 1998, πριν από 12 χρόνια. Τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει ω τμήμα μιας νέας δέσμευσης απέναντι στην Κεντρική Ασία να ολοκληρώσουμε τις εταιρικέ συμφωνίες και συμφωνίες συνεργασίας με όλες τις χώρες και θα πρέπει να αποστείλουμε αντιπροσωπείες σε όλες αυτές τις χώρες, ούτως ώστε να έχουμε μια στεναρή νομική βάση για σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες και να υπάρχει και μια επιχειρησιακή δυνατότητα σε αυτές τις χώρες. Ε, όμως, ε, ακόμη προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις συστάσεις των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Έχουμε επικυρώσει την σχετική συμφωνία με το Τατζικιστάν Έχουμε αναβαθμίσει την, τις αντιπροσωπείες μας σε ορισμένες περιοχές και προσπαθούμε να ανοίξουμε και μια νέα αντιπροσωπεία στο, στη Τασκένδη. Και επίσης, πολύ σύντομα ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε το γραφείο της αντιπροσωπείας μας στην Ασκαμπάντ. Αυτή, είναι αυτές είναι οι πολιτικές ε, που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με βάση τις ε, σχέσεις που έχουμε... Αυτή τη στιγμή μάλλον οι σχέσεις μας με, τα, με το Τουρκμενιστάν είναι περιορισμένες. Βασίζονται στη συμφωνία του 1989 που είναι μιας πρώτης γενιάς ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κοινέ επιτροπέ, τι λεγόμενε κοινή επιτροπή, μία φορά το χρόνο. Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή πριν από δύο-τρει μήνε τέθηκε σε ισχύ, η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία είναι ένα πρώτο θετικό βήμα για να ενδυναμώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Και εδώ μιλάμε για τις εμπορικές ε, διατάξεις της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Και σας ευχαριστώ για την ε, θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009 για αυτή τη συμφωνία. Τώρα, η καινή ώρα για να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για σχέσεις, ε, κάτι το οποίο εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το Τουρκμενιστάν, όπως ακριβώς κάναμε και για άλλες χώρες της περιοχής. Η θέση σε ισχύ της εταιρικής συμφωνίας αυτής θα αντιμετωπίσει πολλά θέματα και θα μας δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής όχι μόνο για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή αλλά και για να προωθήσουμε και τις αξίες μας σε αυτή την πολύ σημαντική χώρα. Μέχρι πρόσφατα, όπως είπε και η κυρία Νικολάη, το Τουρκμενιστάν ήταν μια πολύ κλειστή κοινωνία, μια πολύ κλειστή χώρα και μόνο τώρα, μετά από πολλά χρόνια αυτοαπομόνωσης, ανοίγει ε, και ενώ πέρασε από μια περίοδο δικτατορίας. Ακόμα φέρει τα σημάδια του σοβιετικού παρελθόντος και της ηγεσία του πρώην Προέδρου Νιγιάζοφ. Μετά τις εκλογές ε, του 2007 έχουν αυξηθεί οι συνεργασίες και οι επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από το Τουρκμενιστάν ότι που δείχνει ότι θέλει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για, την, για τις μεταρρυθμίσεις στην, στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, για καλύτερη δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση. Η προσέγγιση της Κομισιόν είναι να έρθουμε σε επαφή, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα, ούτως ώστε να είναι σε καλύτερη θέση για να προωθήσει θετικές εξελίξεις και σε κρίσιμους τομείς, που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέσο δημοκρατίας. Φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μας ανησυχούν πάρα πολύ στη σχέση μας με το Τουρκμενιστάν. Ας μην ξεγελιόμαστε. Το πολιτικό καθεστώς είναι ακόμα αυταρχικό. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι περιθωριακός και τα ΜΜΕ είναι θυμωμένα και ελεγχόμενα. Και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η κυρία Νικολάη αλλά και η κυρία Χέιλ. Αντίθετα από τους προ... τις προλαλήσαντες, προλαλήσασες όμως, πιστεύουμε ότι το Τουρκμενιστάν πρέπει να παίξει το ρόλο του στην διεθνή σκηνή, να κρατήσει την ουδετερότητα και να παίξει ε, το ρόλο του στην περιοχή για τον έλεγχο των συνόρων, την ασφάλεια, τη διαχείριση του νερού, τη χρήση των φυσικών πόρων. Μην ξεχνάτε ότι έχει τους, τα μακρύτερα σύνορα από όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας με το Αφγανιστάν. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες του Τουρκμενιστάν ζητούν στενότερες σχέσεις με άλλους εταίρους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πλήρης ε, και ευρεία αυτή η συμφωνία, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Και για να έχουμε βεβαίως πολιτικό διάλογο τακτικό και για να δημιουργηθεί όλος ο μηχανισμός αυτής της συμφωνίας που σημαίνει ετήσια συμβούλια συνεργασίας, που σημαίνει ε, ετήσια συμβούλια της Επιτροπής που καλύπτουν όλους τους τομείς που μας ενδιαφέρουν και την ε, επιτυχή δημιουργία υποεπιτροπών που μπορούν να συζητήσουν θέματα πολύ ποικίλα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Εμείς βεβαίως συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εξέφρασαν ε, οι ομιλητές για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Αλλά δεν θα πρέπει να αλληλοκατηγορούμεθα μόνο και μόνο γιατί έχουμε διαφορετική οπτική ή διαφορετικές απόψεις. Η κατάσταση είναι άσχημη και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να φτάσουν στο σωστό επίπεδο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Αλλά πιστεύουμε στην Κομισιόν και δεν νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι και το Συμβούλιο το πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες α, επαφής και να έχουμε το σωστό πλαίσιο ε, συνεργασίας με τη χώρα αυτή το συντομότερο δυνατόν. Η κατάσταση θα βελτιωθεί με περισσότερη επαφή, όχι με λιγότερο λιγότερη επαφή. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στα benchmarks, στα ορόσημα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ η ενδιάμεση συμφωνία. Μην ξεχνάμε ότι έχει εφαρμοστεί μόνο από τον Αύγουστο του 2010 και μετά. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις που θέλω να τονίσω. Μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση εν γέννη. Πρώτον, υπάρχει ένα Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που δημιουργήθηκε, ε, που έχει σημαντικούς πόρους, που το καθήκον του είναι να βοηθάει το Τουρκμενιστάν να εφαρμόσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ε, περάσει τις απαραίτητες ε, αλλαγές ε, στην εσωτερική νομοθεσία. Υπάρχει ένα διαμεσοβελαβητής. Υπάρχει ένας επίτροπος, κρατικός επίτροπος για να εξετάζει αιτήματα πολιτών για την εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν εκεί. Ένας νέος ποινικό κώδικας υιοθετήθηκε το Μάιο, ε, μειώνοντας ε, την μέγιστη ποινή φυλάκισης για τα σοβαρά εγκλήματα και μεταρρυθμίζοντας το σύστημα καταδίκης και τιμωριών, δηλαδή προτάσσονται τώρα, προτιμώνται τώρα τα πρόστιμα και όχι οι φυλακίσει. Αυτέ είναι οι τρεις βασικές εξελίξεις που ήθελα να τονίσω. Επίσης, ε, ε, έχουμε συζητήσει κάτι επανάληψη λεπτομερώς με τις αρχές στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, κυρίως έχουμε συζητήσει το θέμα των περιορισμών για τους ταξιδιώτες, οι οποίοι οι περιορισμοί έχουν μειωθεί, ε, έχει διευκολυνθεί η κίνηση στα σύνορα με την κατάρτιση των εσωτερικών ελέγχων. Όμως υπάρχουν ακόμα πολύ σημαντικοί περιορισμοί για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η Κομισιόν έχει θέσει το θέμα αυτό στις Τουρκμενικές Αρχές και ιδίως το θέμα του μαυροπίνακα ε, όπου αναγράφονται τα άτομα τα οποία δεν επιτρέπεται να βγουν από τη χώρα. Αυτό μας ανισχύει πάρα πολύ. Το δεύτερο σημείο είναι η πρόσβαση στις φυλακές για το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε, το θέμα, έχουμε θέσει το θέμα αυτό κατ' επανάληψη στις αρχές. Είναι κάτι που μας ανησυχεί και για άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας, αλλά και έχει σημειωθεί περισσότερη πρόοδος. Οι φυλακές του Τουρκμενιστάν είναι κλειστές σε διεθνείς παρατηρητές. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δυνατότητα παρατηρητών. Ε, γίνονται επαφές μεταξύ των αρχών του Τουρκμενιστάν και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι δίνουμε βοήθεια για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξελίξει για να βοηθήσει το Τουρκμενιστάν να αναπτύξει το δυναμικό εγχώρια για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα με 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία και στα πλαίσια του μέσου ε, εκδημοκρατισμού και πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια πρώτη προσπάθεια σοβαρή από πλευρά του Τουρκμενιστάν. Υπάρχουν και άλλα ε, μικρότερα προγράμματα ε, για τα ΜΜΕ με τη συμμετοχή και του BBC και την δημιουργία ε, δυναμικού διακυβέρνηση. Στην Άσκαμπα έχουμε μια νέα αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει για την σοβαρή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Δεν έχουμε αυταπάτε. έτσι, έτσι κλείνω, έτσι καταλήγω. Δεν είναι ιδανική η κατάσταση σε καμία περίπτωση, αλλά Νομίζουμε ότι η μη ανάμειξη δεν είναι σωστή δυνατότητα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω για τι τελευταίε αυτέ πληροφορίε, για τι ε, συγκεκριμένε <clears throat> βελτιώσει που έχουν έρθει στη γνώση του και φυσικά για το δρόμο που παραμένει να διατρέξουμε. Θα ήθελα να δώσω τώρα στην Αντρέα Μπέρκ, η οποία εκπροσωπεί το Human Rights Watch, που είναι ιδιαίτερα ενεργό στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίε καθώ και κύριοι. Όπως έχει λεχθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιζητεί αναβάθμιση των σχέσεών της με το Τουρκμενιστάν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει πλήρως τη δυνατότητά της να δράσει ως καταλήτης για θετική αλλαγή στο Τουρκμενιστάν. Η πεποίθησή μα είναι ότι θα πρέπει να τονίσει και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις ανησυχίες του και να υπενθυμίσει στην Κομισιόν και το Συμβούλιο την υπόσχεσή τους να αγοριστούν για ουσιαστική αλλαγή και βελτίωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από την εφαρμογή της εταιρική συμφωνίας και συμφωνίας συνεργασίας. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτής της συμφωνίας θεώρησε ότι παραθέτω, είναι ένα μοχλό πίεση για να ενισχυθεί η δημοκρατική μεταρρύθμιση στο Τουρκμενιστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα θα πρέπει να εξετάσει μια πλήρη συνεργασία και εταιρική σχέση με το Τουρκμενιστάν. Είναι όμω τώρα σε αυτή τη φάση πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια σοβαρή και ειλικρινή αξιολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων που είχε η εταιρική σχέση με το Τουρκμενιστάν, αν υπήρξαν τέτοια αποτελέσματα και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναβάθμιση θα εξαρτάται από περαιτέρω βελτιώσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επειδή αναφερθήκανε οι βαθμονομήσει στα benchmark διάφορε φορέ, θέλω να τονίσω για ορισμένα από αυτά τα στοιχεία <clears throat> αξιολόγησης και την πρόοδο ή μη πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Καταρχήν, ένα τέτοιο πρώτο κριτήριο, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, ήταν η χωρίς όρους χωρις όρου όλων των ε, πολιτικών κρατουμένων. Ένας άγνωστο αριθμός τέτοιων ατόμων βρίσκεται ακόμα στις φυλακές με κατηγορίες οι οποίες έχουν, από ό,τι φαίνεται, πολιτικά, πολιτικά κίνητρα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δίωξη και οι δίκες και η απουσία ξένων παρατηρητών δεν μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε ένα αξιόπιστο αριθμό για τους πολιτικούς κρατουμένους, να εξασφαλιστεί ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των κατηγοριών εναντίον του. Τα τελευταία χρόνια ήταν ακόμα πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του ποινικού συστήματος για πολιτικούς στόχους, γιατί όλο και λιγότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης του Τουρκμενιστάν για την φυλάκιση <clears throat> ατόμων με υψηλό προφίλ. Τέτοιοι είναι ο Μαλκουρμπάν, Κίτσεφ, Σαπαρτουρντή, Χότζεφ, οι οποίοι έχουν εργαστεί σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο Γκουγκέλτη Ανανιάζοφ, ο πολιτικός αυτός αντιφρονούν, αντιφρονούντας. Μετά από τον θάνατο του κυρίου Νιάζοφ, που ήταν Ισόβιος πρόεδρος το 2006, η κυβέρνηση απελευθέρωσε ορισμένου πολιτικού κρατουμένου. Αλλά έκτοτε η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν όχι μόνο είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για την αναθεώρηση, για την αναψηλάφιση μάλλον των υποθέσεων που έχουν οδηγήσει σε φυλάκιση και να απελευθερώσει αυτού οι οποίοι έχουν άνομα φυλακιστεί, δεν έχει καν αναγνωρίσει ότι το θέμα των πολιτικών κρατουμένων είναι μια σημαντική πτυχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη αποτυχία τη κυβέρνηση είναι το γεγονό ότι δεν δέχτηκε ουδεμία από τι συστάσει που έγιναν για το θέμα αυτό μέσα στη, στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη επισκόπηση μάλλον του Τουρκμενιστάν το 2008 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ένα δεύτερο κριτήριο, benchmark, αφορούσε την άρση όλων των εμποδίων για την ελεύθερη μετακίνηση. Ενώ κάποιοι ακτιβιστές είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, οι αρχές του Τουρκμενιστάν αυθαίρετα εμποδίσουν <clears throat> πολίτες τους να πάνε στο εξωτερικό και μετά να γυρίσουν βάσου, βάσει ενός αυθαίρετου συστήματος απαγόρευσης ταξιδίου που αφορά τους αντιφρονούντες και τους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Σφεντλάνα Σοράσεβα, η αδερφή μιας εξορία ηγέτηδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπόκειται σε απαγόρευση ε, ταξιδίου, όπως και ο άντρα τη, ο οποίο δεν μπόρεσε να τύχει ιατρική περίθαλψη και πέθανε. Ελήψη τέτοια περίθαλψη. Το 2009 αυξήθηκαν οι περιορισμοί με μια νέα απαγόρευση ταξιδίου που αφορά τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάνε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως στο Κυργιστάν. Ενώ στο παρελθόν μπορούσαν πολλοί φοιτητέ να φοιτούν σε γειτονικέ χώρε συγκεκριμένα στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ασίας, εκεί οι φοιτητέ οι οποίοι θέλουν να πάνε εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν επίση για θρησκευτικού στόχου είναι στόχοι αυτών των περιορισμών. Το τρίτο κριτήριο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η πρόσβαση για εξωτερικούς ανεξάρτητους παρατηρητές και αναφέρθηκε εδώ το θέμα των παρατηρητών του Διεθνούς Εθνικού Σταυρού. Κανένας εξωτερικός φορέας δεν έχει μπορέσει να ερευνήσει τα θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στη χώρα αυτή και κανένας φορέας κυβερνητικός ή μη κυβερνητικός έχει πρόσβαση στα σοφρονιστικά καταστήματα και στους χώρους κράτηση Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση για ανεξάρτητους παρατηρητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Εννέα τέτοιες αποστολές του ΟΗΕ δεν μπόρεσαν να πάνε, επίσης αποστολές του Ερυθρού Σταυρού και άλλων φορέων. Το Σεπτέμβριο του 2008 ο ειδικό εισηγητής για την ελευθερία θρησκείας επισκέφθηκε τη χώρα και αυτό έδωσε λαβή σε ελπίδες ότι θα ακολουθήσει ένα πιο ανοιχτό πνεύμα στη χώρα αυτή για την ανεξάρτητη παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά μετά από δύο χρόνια είναι σαφές ότι δεν υπήρξε καμία συνέχεια και το Τουρκμενιστάν παραμένει ερμητικά κλειστό σε οποιαδήποτε μορφή εξωτερικού ελέγχου. Η Jacqueline Hale αναφέρθηκε ήδη στην κατάσταση των Medicine Sans Frontier, των ιατρών χωρίς σύνορα, που αναγκαστήκανε τον Δεκέμβριο του 2009 να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ένα άλλο κριτήριο ήταν η βελτίωση των αστικών ελευθεριών το δικαίωμα ελευθερίας του συνεταιρίζεσθε και το δικαίωμα ελευθερίας της, η ελευθερία της έκφρασης, στο Τουρκμενιστάν οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές δεν μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και στο Τουρκμενιστάν και εν εξορία εξακολουθούν να παραμένουν σε συνεχή παρακολούθηση και με το φόβο συνεχών αντιπίνων από την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν. Τον Οκτώβριο εφέτος 2010 οι εξωματούχοι του Τουρκμεν Νιστάν προσπάθησαν να εμποδίσουν ακτιβιστές να συμμετάσχουν στην ε, συνδιάσκεψη επισκόπησης της ΟΑΣΕ στην Βαρσοβία. Και αναφέρθηκε ήδη και η κυρία Πρόεδρος για τον, στον κύριο Τούχ Πατουλίν, ο οποίος βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση. Οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν τους ακτιβιστές να μην συναντούν εκπροσώπους του ΟΗΕ και άλλων φορέων, ούτε καν τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ, την εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα θέματα ελευθερίας θρησκείας, θρησκευτική έκφρασης. Κανένας διεθνής εισηγητής δεν μπόρεσε να μπει στο Τουρκμενιστάν το τελευταίο καιρό. Ο νόμος περί συνεταιρίζεστε έχει τύχει επίκρισης γιατί θέτει ε, ανεδαφικές απαιτήσει μη ρεαλιστικέ απαιτήσει για μη κυβερνητικέ οργανώσει για να καταγραφούν στα Μητρώα. Ζητάει να έχει, παραδείγματο 500 μέλη ένα τέτοιο φορέα. Υπάρχει απόλυτη, απόλυτη έλλειψη ελευθερία έκφραση. Τα έντυπα μέσα και η τηλεόραση ελέγχονται απόλυτα από την κυβέρνηση. Είναι πολύ δύσκολο για τα μέσα ε, ενημέρωση να έχουν ανταποκριτέ στο Τουρκμενιστάν γιατί και οι ανταποκριτές τους και οι δημοσιογράφοι ελεύθεροι που συνεργάζονται με αυτούς έχουν ξυλοκοπηθεί και τρομοκρατηθεί. Εμποδίζεται η πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν μπορεί να πάει κανείς σε ένα ίντερνετ καφέ χωρίς να δείξει το διαβατήριό του και η κυβέρνηση παρακολουθεί πλήρω όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση σε ξένες εφημερίδες ή περιοδικά γιατί όλα αυτά τα κατάσχουν οι συνοριακοί φρουροί στην είσοδο στη χώρα. Μόνο έντυπα μέσα τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο Τουρκμενιστάν. Μπορεί κανείς να διαβάσει εκεί. Κλείνω και με την ε, ανάγκη να υπάρξει μεταρρύθμιση σε όλους τους φορείς και σε όλα τα επίπεδα της ε, κρατικής μηχανής. Το 2010 το Τουρκμενιστάν ενέκρινε μία σειρά νόμων που τροποποιούν και τον ποινικό κώδικα και τον διοικητικό κώδικα και τα, τον κώδικα για την άσκηση του Επαγγελματό του δικηγόρου. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δημόσια λογοδοσία τη κυβέρνηση. το Τουρκμενιστάν έχει μία ενιαία μορφή εξουσία. Ο πρόεδρος είπε ότι είχε πει πρόσφατα ότι είναι έτοιμη η χώρα για μία πολυκομματική πολιτική ζωή, αλλά ακόμα δεν έχει ε, εγκριθεί η λειτουργία οποιοδήποτε ανεξάρτητου πολιτικού κόμματος. Με το νέο σύνταγμα το 2000, του 2008 ο πρώτος μπορεί να διορίζει και να απολύει δικαστικούς χωρίς έλεγχο από το Κοινοβούλιο, δημιουργεί την εκλογική επιστροπή, επιτροπή και μπορεί να ε, δημοσιεύει διατάγματα χωρίς κανένα έλεγχο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο, ούτε καν διαμεσολαβητής. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έδωσε το πράσινο φως στην ενδιάμεση εμπορική συμφωνία ανέμενε δε θετικά αποτελέσματα από αυτήν την διαδικασία. Εφόσον όμω δεν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναστείλει την υποστήριξή του για το επόμενο βήμα, δηλαδή την εταιρική συμφωνία και συμφωνία συνεργασία, μέχρι ότι το Τουρκμενιστάν κάνει όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεών μα με την όμορφη αυτή χώρα. Σα ευχαριστώ, κύριε Μπέργκ. Άρβινσον από το γραφείο του ΙΠΑ του Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών, η επόμενη ομιλήτρια. Ίσως να αλλάξετε θέση για να μιλάτε μπροστά στο μικρόφωνο. Thank Ευχαριστώ. Πάρα πολλά ουσιαστικά θέματα έχουν ήδη αναφερθεί από όλους τους ομιλητές για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Δεν θα επισέλθω λοιπόν και εγώ σε περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη στο Τουρκμενιστάν τα τελευταία χρόνια μετά από το άνοιγμα προς τα έξω της χώρας που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια. Το Μάιο του 2007 ο πρώην υπατοσαρμοστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κυρία Αρμπόρη ήταν η πρώτη ε, επίτροπος που επισκέφθηκε το Τουρκμενιστάν. Υπογράμμισε τότε ότι η σημασία της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και την παροχή δημοκρατικής ελευθερίας για την άσκηση των δραστηριοτήτων και η εξασφάλιση σωστή σωστής ανάμεσα στα εστρία ε, όργανα της εξουσίας και η δημιουργία ενός πραγματικά ε, ανεξάρτητου Ινστιτούτου, Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με τι αρχέ του Παρισιού ήταν προτεραιότητε που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα. Ο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπαν Κιμούν, στι αρχέ Απριλίου φέτο επισκέφθηκε το Τουρκμενιστάν και είχε την ευκαιρία να αισθανθεί με τον Πρόεδρο και με τον Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Δημοκρατία και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να συζητήσει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αυτού του φορεί κατά την διάρκεια τη επίσκεψή του ως γραφείο ε, τον Ιούνιο του 2008 το Κυργιστάν και το γραφείο του είπα του Επιτρόπου υπέγραψαν μια συμφωνία για τη δημιουργία του γραφείου που εξυπηρετεί το Τουρκμενιστάν, το Κυργιστάν και το Τουρκμενιστάν και υπάρχουν και ομάδες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ύπατη αρμοστία και του UNDP, το, αναπτυξιακό, το πρόγραμμα, ε, ε, ε, αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ, συνεργάζονται για να σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας και της ικανότητας των κατοίκων του Τουρκμενιστάν να έρχονται σε επαφή με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Εκπαιδεύομαι αξιωματούχους κρατικούς λειτουργούς του Τουρκμενιστάν ε, από διάφορες διοικητικές υπηρεσίες για την υποχρέωση τήρησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος παρέχουμε πληροφορίες ε, ε, για, το, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προγράμματα ευαισθητοποίησης και στις πέντε επαρχίες. Αυτή η διαδικασία άρχισε σχετικά πρόσφατα και αυτό που ελπίζουμε είναι ότι η υλοποίηση, η εφαρμογή ε, των ε, συστάσεων θα προχωρήσει περισσότερο από ό,τι σήμερα, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές ε, για τους ανθρώπους, για τους κατοίκους της χώρας. Σε ό,τι αφορά την οικουμενική περιοδική επισκόπηση του Τουρκμενιστάν ήταν η πρώτη χώρα που υπέστη αυτή την επισκόπηση το 2008 και τις υποβλήθηκαν συστάσεις για την κατάργηση των βασανιστήριων, την ελευθερία θρησκείας, ελευθερία κυκλοφορίας, ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για να αναφέρουμε τις πιο σημαντικές συστάσεις που είχε δεχθεί τότε το Τουρκμενιστάν. Απέριψε όμως και άλλες σημαντικές συστάσεις συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για την απαγόρευση του ταξιδιού, την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και για την αναθεώρηση περιπτώσεων κρατουμένων για πολιτικούς λόγους. Όπως αναφέρθηκε επίσης με σε μια θετική προσπάθεια δέχθηκε τον ειδικό εισηγητή για την ελευθερία ε, της θρησκείας που επισκέφθηκε τη χώρα το 2008. Ήταν η πρώτη επίσκεπτη ενός εισηγητή στο Τουρκμενιστάν. Αλλά ε, νέα άλλοι έχουν υποβληθεί διάφορες ε, προτάσεις για επισκέψεις από τον εισηγητή για την εξαρτησία των δικαστών και νομικών τον εισηγητή για τα βασανιστήρια, τον εισηγητή για τις εξοδικαστικές εξελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, τον εισηγητή για τις ε, κρατήσεις, το εισηγητή για το δικαίωμα στην παιδεία. Επίσης ζήτησε να επισκεφθεί τη χώρα και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση για να γίνει αυτή η επίσκεψη του χρόνου, αλλά δεν έχει τίποτα ακόμα επιβεβαιωθεί. Τέλος, για τα μέσα ε, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά το άνοιγμα της χώρας έχουν γίνει κάποιες θετικέ κινήσεις, παραδείγματο χάρη σύμβαση για το δικαίωμα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, ε, υπεγράφει, επικυρώθηκε πρόσφατα, αλλά υπάρχουν άλλα διεθνή κείμενα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν έχουν επικυρωθεί από τη χώρα όπως το πρωτόκολλο στη σύμβαση κατα, ε, των βασανιστήριων που, θα, που προβλέπει επισκέψεις και ελέγχους στα κέντρα κράτησης. Αυτά συνοψίζοντας αυτό που συνοψίζω θα ήθελα να πω, αυτό που έχει σημασία είναι να, να να συνεχιστεί η παρακολούθηση αυτής της χώρας και ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε θα έχει πολύ θετικέ επιπτώσεις για το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστώ. Και τώρα ας πέρασουμε στη συζήτηση. Δύο άτομα ζητάνε προς το παρόν το λόγο. Ο κύριος ε, Σίβιετς και ο κύριος Γκζίμπ. Ο κ. πρώτος. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τους ομιλητές. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε πράγματα για το Τουρκμενιστάν ε, έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα. Θυμάμαι μια πρώτη συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, όταν είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε την έκθεση. Και πρέπει να ομολογήσω ότι τα όσα γνώριζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πραγματικότητα του Τουρκμενιστάν ήταν ανεπαρκή ξεπερασμένα. Άκουσα και εκτίμησα τα όσα μας είπαν οι ομιλητές ε, σήμερα, γιατί οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι φορείς που ασχολούνται με αυτά, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Τα ακούσαμε αυτά και στην έκθεση που μας παρουσιάστηκε σήμερα όλες τις χώρες πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Όλες τις χώρες πρέπει να τις εξετάζουμε. Ε, δεν πρέπει να παραμαλούμε καμία χώρα, κανένα πολίτη καμίας χώρας. Ακόμη και ένα άτομο αν υποφέρει είναι αρκετό, είναι υπερβολικό. Έχουμε ένα κατάλογο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και από την άλλη έχουμε αυτούς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε τους καλούς και τους κακούς. Ε, και από την άλλη έχουμε την άλλη νομίσματος την επικύρωση της ε, συμφωνίας αυτής με το Τουρκμενιστάν. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των διαφόρων οργανώσεων και φορέων και θέλω να τους πω ότι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άτομο το οποίο είναι αμεληταίο. Όλοι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, όλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα ή να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ε, δεν μπορεί να φυλακίζεται κανένα γιατί δεν θέλει να εκτίσει την ε, στρατιωτική, να εκτελέσει τη στρατιωτική του θητεία. Όχι, στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε. Μαζί σα είμαστε. Ε, και μάλιστα έχω την εντύπωση ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μαζί μα. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προασπίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένω, εδώ αντιμετωπίζω ένα ψεύτο δίλημα στην πραγματικότητα. Έτσι νομίζω. Το αν θέλουμε δηλαδή να υπερασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Όχι, προφανώ και θέλουμε. Το βασικό δίλημα είναι πώ θα δημιουργήσουμε σχέσει με τη χώρα αυτή, με το Τουρκμενιστάν, ούτω ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω ώστε να έχουμε πολύ άριθμε επαφές με το Τουρκμενιστάν. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και όχι αν θα το κάνουμε αυτό, αν θα έχουμε επαφές δηλαδή. Ε, το πώς θα το κάνουμε μπορεί να απαντηθεί ως εξή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παλιά νομικά εργαλεία της Σοβιετικής εποχής, γιατί αυτή η συμφωνία υπογράφτηκε με την τότε ε, Σοβιετική Ένωση που δεν υπάρχει σήμερα και παρατάθηκε η ισχύ για να ισχύσει για τις σημερινές χώρες που προέκυψαν από τις τάχτες της Σοβιετικής Ένωσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το απαρχαιωμένο εργαλείο ή χρειαζόμαστε κάτι το καινούριο. Αυτό υπογράφηκε πριν από 12 χρόνια. Και είναι πολύ περίεργο να έχουμε μια συμφωνία που υπογράφτηκε 12 χρόνια πριν και να, χρειαστούν, να, να χρειαστεί να περάσουν 12 χρόνια για να επικυρωθεί μια τέτοια συμφωνία. Αυτό είναι περίεργο. Θέλω να ξεπεράσουμε τα συναισθήματά μας και να μιλήσουμε για την πολιτική. Γιατί αν μπλέξουμε με τα συναισθήματα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά μετά και να βρούμε αποτελεσματικά εργαλεία για να προωθήσουμε πολιτικές. Επί τρεις γενιές στο Τουρκμενιστάν ήταν υπό, τον κομμουνιστικό, υπό την κομμουνιστική εξουσία. Ε, όσοι έζησαν σε τέτοιε χώρε γνωρίζουν πώ ε, λειτουργούσε ο κομμουνισμό, ο οποίο αδιαφορούσε, για να το πω ήπια, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Τουρκμενιστάν επιπλέον αντιμετώπιζε την πραγματικότητα μιας ασιατικής χώρας. Αν εμένα μου κάνει την ερώτηση, αν θα προτιμούσα να ζήσω τον κομμουνισμό τη Πολωνία, τον κομμουνισμό του Τουρκμενιστάν, ε, θα έλεγα καλύτερο ο κομμουνισμός τη Πολωνία. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν για τρει γενιέ τον κομμουνισμό. Δηλαδή, αυτό που ενηλικιώθηκε το 1990 δεν είχε ένα παππού που θα μπορούσε, που θα μπορούσε να του πει πώ ήταν η ζωή πριν τον κομμουνισμό. Επομένως, η ιστορική κατάσταση είναι δύσκολη. Η νοοτροπία της κοινωνίας έχει επηρεαστεί από την ιστορία της χώρας αυτής. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γιατί μην ξεχνάμε πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες σε μια κοινωνία στους στην ομάδα των σοσιαλιστών συζητάμε αυτό το θέμα, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας. Η σημερινή ακρόαση είναι πολύ σημαντική γιατί μας κάνει να συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει στη χώρα αυτή. Χαίρομαι που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση και θέλω να επαναλάβω το εξή. Ας αποφύγουμε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως Κοινοβούλιο να κάνουμε τίποτα. Χρειάστηκαν 12 χρόνια για να προχωρήσουμε. Ας ηρεμήσουμε και ας δούμε τι απόφαση θα πάρουμε. για αυτή τη συμφωνία. Κάθε μήνα ασχολούμαστε ε, με το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν συνεδριάζομαι στο Στρασβούργο. Δεν νομίζω ότι συζητήσαμε ούτε μία φορά παρόλα αυτά το Τουρκμενιστάν. Είναι μία παράληψη νομίζω. Ο κύριος Γκζίμπ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε μια σημαντική απόφαση και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε σύγκρουση δύο αντιμαχόμενων, αντιμαχόμενων θέσεων. Η μία θέση θεωρεί ότι ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια συνθήκη η οποία έχει κυρωθεί και μας ε, θέτουν το ερώτημα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα ώστε να μπορούμε να αναβαθμίσουμε τι τις σχέσεις μας. Και βλέπουμε τώρα όλα αυτά τα προβλήματα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ αυτό το εγχείρημα, αυτή η εφαρμογή της συμφωνίας. Θα επανέλθω και σε αυτό που είπε η κυρία Νικολάη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά από το 2008 και 2009, είχε θεσπίσει ορισμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να εκπληρωθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δυστυχώ πρέπει να πούμε απερίφραστα ότι δεν εκπληρώθηκαν αυτά τα κριτήρια από την πλευρά του Τουρκμενιστάν. Εμεί δεχτήκαμε την ενδιάμεση συμφωνία, αλλά τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να πράξουμε σε, στις ε, σημερινές Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια συμφωνία εταιρικού χαρακτήρα και συνεργασίες. Έχουν παρουσιαστεί επιχειρήματα από τους ε, εισηγητές μας. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το σύνολο όλων αυτών των θεμάτων, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε κάποιο από αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά αυτά που είπε και ο κύριο Βίγκαντ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά είναι σημαντικά επιχειρήματα. Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει οποιαδήποτε διαδικασία σε μια χώρα όπου δεν υπάρχουν εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αναβαθμίσουμε λοιπόν τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή, αυτό θα έχει το θετικό αποτέλεσμα ότι θα έχουμε εκπροσώπους θα αναπτύξουμε μηχανισμούς που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε περιοδικά εκτίμηση της αλλαγής της κατάστασης του Τουρκμενιστάν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Για το αν επιτυγχάνεται η τήρηση των benchmarks, των κριτηρίων, για το αν υπάρχει μία βελτίωση ή μία επιδείνωση της κατάστασης και στην περίπτωση που δεν εκπληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως την λειτουργία αυτής της συμφωνίας. Ούτως εμείς ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε να κάνουμε μια επιλογή. Εγώ χαίρομαι που η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχει ακόμα πάρει την τελική της απόφαση πρωτού εμείς ως Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η Ευχαριστώ τον κύριο Αντιπρόεδρο για τη θαυμάσια ανάλυση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. <clears throat> Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Ντόμσκι τώρα να λάβει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Απλώ μερικέ ε, σύντομε παρατηρήσει. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε κοινοτοπίε, κλισέ και συγκινησιακέ αντιμετωπίσει για χώρε όπω το Τουρκμενιστάν. Ένα πράγμα είναι απόλυτα σίγουρο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα επί τόπου. Δεν μπορούμε να μπλεχτούμε σε ένα ευχολόγιο και σε μία σειρά ευσεβών πόθων που λέμε ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα και να τα θεωρήσουμε αυτά σε δεδομένα. Θα πρέπει να βασιστούμε στα πραγματικά γεγονότα. Από τη μία πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να έχουμε επαφή με το Τουρκμενιστάν, να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγχρόνω όμω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν θεσμοί με του οποίου να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το απτό για να μπορέσει να υπάρξει συνεργασία. Αν δεν έχουμε εργαλεία για την παρακολούθηση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι υποκρύπτεται ε, ανάμεσα στις λεπτομέρειες ο διάβολος και πολλές φορές η συνεργασία και η επαφή μπορεί να βοηθήσουν μια κοινωνία η οποία έχει απομονωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ίσως με λανθασμένες <clears throat> ενέργειες από τη δική μας πλευρά μπορεί το καθεστώς εκεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι ένα σήμα αποδοχής, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να επισημοποιήσουμε κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά ένα δίλημα. Αυτό το οποίο θέλουμε όλοι είναι να ασκήσουμε πίεση για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε όμως τα εργαλεία και τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό ή όχι. Ευχαριστώ. Τα ευχολόγια δεν βοηθάνε. Νομίζω ότι πρέπει να σας ακούσουμε και νομίζω ότι και η συγγήτρια σκέφτεται με ποιους μηχανισμούς μπορούμε σε περίπτωση που αυτή η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας επικυρωθεί, να μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, να έχουμε κάποιους μοχλούς, να έχουμε κάποιους μηχανισμούς. Ε, όταν επικυρώσαμε την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία, λειτουργήσαμε με ευχολόγια ως Κοινοβούλιο. Άκουσα πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Δεν είναι ευχάριστο να ακούμε πως ε, τα benchmark, τα δικά μας, δεν υλοποιήθηκαν Επουδενή, σε καμία περίπτωση. Αν προχωρήσουμε λοιπόν, χρειαζόμαστε μια βάση για να προχωρήσουμε. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο και η Υποεπιτροπή ε, δεν έχουν αποστρέψει το βλέμμα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να εμπλακούμε μέσα στα όρια που προβλέπονται, τα νομικά όρια. Προσπαθώ να καταλάβω την ε, διαφορά της ε, νομικής βάσης, της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας και αυτής της ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσπαθώ να δω διαφορά, δεν βλέπω διαφορά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μας πει η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου ποια είναι η βάση, ποια είναι η διαφορά. Α, δεν είναι παρούσα η νομική υπηρεσία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε στην νομική υπηρεσία για να μας διαφωτίσει για το θέμα της νομικής βάσης και για να διερευνήσουμε το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης. Η συγγήτρια το έχει υπόψη της αυτό. Αυτές είναι δικές μου προσωπικές ε, σκέψεις, ακούγοντας τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και των εμπειρογνωμών. Αλλά καιρός να επιστρέψουμε ξανά στην εισηγήτρια για να μας απαντήσει. Ο κύριος Ομπιόλς. Για αυτή την έλλειψη μηχανισμού σχέσεων, ε, ελέγχου. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει δυνατότητα βραχυπρόθεσμα να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του Κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν. Αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Δεν έχω καμία πληροφορία. Δεν ξέρω αν εσεί, Πρόεδρε, ή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουν κάποιε πληροφορίες, αν μπορούν να μας πούν κάτι για αυτό το θέμα. Κύριο Μπιόλς. Ας ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Νικολάη, ε, και μετά θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για αυτή τη σημερινή συνεδρίαση, γιατί νομίζω ότι χύνει το φως στο τι συμβαίνει στο Τουρκμενιστάν. Όλοι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο, όλοι τα ίδια θέλουμε. Όλοι θέλουμε να έχουμε συμφωνίες συνεργασίας, που θα οδηγήσουν σε κάποιες αλλαγές στη χώρα. Εν προκειμένου μας απασχολεί το Τουρκμενιστάν. Θέλουμε να έχουμε συμφωνίες συνεργασίες, αποτελεσματικές. Μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στη βελτίωση της κατάστασης του Τουρκμενιστάν. Ο κύριος Ντάνσκης έχει κάποιες αμφιβολίες. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά το ρόλο των ε, ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετά την ε, ένταξή τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξέχασαν ότι τα πρότυπα τα οποία επιβάλλονται θα πρέπει να υλοποιούνται κιόλας και η δική μου χώρα είναι ένοχη σε αυτό. Το θέμα είναι τι στάση έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι σε αυτές τις συμφωνίες. Νομίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να, προωθηθούν, να προωθούνται ούτω ή άλλω. και να τα προασπιζόμαστε ούτω ή άλλω. Αλλά πώς. Κοιτώντα με το κι άλλη μια μακρινή χώρα ή προσπαθώντας να κάνουμε κάτι. Εγώ είμαι ανοιχτή και ευχαριστώ τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές για τις προτάσεις τους. Περιμένω και τροπολογίες γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε τροπολογίες. Θέλω να συνεργαστούμε για να βρούμε συνεπείς ε, μηχανισμούς, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι η θέληση των ευρωπαϊκών λαών, να γίνει σεβαστή σε όλες τις συμφωνίες. Προτιμώ να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία όμως να έχουν βάση και όχι τυπικά, τυπικότητες. Νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιτρέπει να εμπλακούμε και να ξεπεράσουμε τις τυπικότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Να σας απαντήσω κύριο Μπιόλς. Τον Ιούλιο έγραψα στον το ε, πρόσωπο και στους συναδέλφους για τη σημασία της επερχόμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Στις 6 Αυγούστου μου απάντησε ο ύπατος εκπρόσωπος. Βρίσκεται στο φάκελο, αλλά τον ξαναβρή, την ξαναβρήκα αυτήν την επιστολή. Κοιτάξτε τι κι εσείς. Λοιπόν, για το ερώτημά σας, ε, κυρία Ομπιόλς. Η κυρία Άστον αναφέρεται στην πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη χωρίση βοήθεια του Τουρκμενιστάν και στην πρόθεση να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ε, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και του εξυγχρονισμού του Κοινοβουλίου. Με τη βοήθεια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που με εξέπληξε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι είπα εκπρόσωπος μου γράφει ότι απουσία μιας ε, επικαιροποιημένης νομικής βάσης με δεσμευτική αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, περιοριζόμαστε. Ε, δεν βλέπω να υπάρχει καμία διαφορά με την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία στη νομική βάση. Η ύπατη εκπρόσωπο πιστεύει ότι η δέσμευσή μα απέναντι στο Τουρκμενιστάν ε, σε ό,τι αφορά και τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να ενδυναμωθεί εφόσον τεθεί σε ισχύ αυτή η εταιρική συμφωνία και όταν υπάρξει αυτή η αντιπροσωπεία μας στην Άσκαμπα. Ε, υπάρχουν διαφορετικές λύσεις από ό,τι άκουσα στις α, ε, διαφορετικές ασιατικές χώρες. Και διαφορετικές προϋποθέσεις για το Τατζικιστάν, ε, το Τουρκμενιστάν, υπό τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπεία, να εγκατασταθεί μια αντιπροσωπεία. Επομένως, η επικύρωση αυτής της συμφωνίας δεν είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές. Επίσης γράφει, είπα την εκπρόσωπος, ότι αυτή η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα μας δώσει μια περαιτέρω νομική βάση για περαιτέρω σχέσεις και διάλογο, αλλά θα μας δώσει και ένα εργαλείο για διμερείς σχέσεις ε, με σκοπό ε, την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και σε άλλες τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει παρόμοιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συμπεριλαμβανομένων εδώ και όλων των υπολείπων χωρών της, της α, Κεντρικής Ασίας. Ποια είναι η νέα αυτή νομική βάση, μπορείτε να μου εξηγήσετε και αυτές οι δεσμευτικές αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι εδώ. Μπορεί να μας απαντήσει λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που είπε η Επιτροπή στη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της ενδιάμεσης συμφωνίας που σημαίνει ότι υπάρχει ότι έχουν τα, τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο αυτής της ε, συμφωνίας που μεταφέρθηκε στην ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με ακριβώς την ίδια διατύπωση στο άρθρο 1 στη μελλοντική ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στο άρθρο 2 με βάση το, και στο, ε, στο άρθρο 28 και 98 των δύο συμφωνιών αντίστοιχα που αναφέρονται σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχει κοινή διακήρυξη από τις δύο πλευρές που ε, ε, αναφέρεται συγκεκριμένα στο γεγονός ότι αυτά αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία στο άρθρο 1 της ενδιάμεσης συμφωνίας ή στο αντίστοιχο άρθρο της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Η διατύπωση της συμφωνιας εταιρικη σχεση και συνεργασιας πολύ σωστά το είπατε, και στα δύο κείμενα. Αλλά η κάλυψη της δεύτερης συμφωνίας είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει ασφαλώς πολλούς περισσότερους τομείς τους οποίους θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε δράσεις με το Τουρκμενιστάν, προβλέπει τον πολιτικό διάλογο για τα θέματα αυτά και προβλέπει μια ειδική θεσμική δομή για την πρόθεση των πολιτικών και της στρατηγικής μας. Και υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης, προβλέπεται επίσης μια διαδικασία παρακολούθησης των σχέσεων με το Τουρκμενιστάν. Πιστεύουμε λοιπόν ακράδαντα ότι η ευρύτερη νομική βάση θα μας δώσει μεγαλύτερο, ευρύτερη κάλυψη και πιο πολλές θεσμικές δυνατότητες για να παρακολουθούμε πιο αποτελεσματικά τις εξελίξει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι εκτι... αντιλαμβάνομαι αυτά που είπε ο ενοπληρωτής πρόεδρος και ο κ. Στεβίνσκι, ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε ένα ψευδοδήλημα. Δεν είναι ε, για, τους, για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ποια μέσα, ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε για να εξασφαλίσουμε ε, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και εκεί μπορεί να υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ μας και εγώ σας παρουσίασα, ελπίζω με σαφήνεια, τη θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου και που είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο λαός του Τουρκμενιστάν θα το ερμήνευε σαν κακό μήνυμα εάν η απόφαση είναι ότι δεν θέλουμε ε, να έχουμε με σας μια συμφωνία αντίστοιχη με εκείνη που έχουμε υπογράψει με τις γειτονικές σας χώρες τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο τα πρότυπα του Τουρκμενιστάν όπως έχουν γίνει και πρότυπα των υπόλοιπων χωρών της περιοχής με τη συμφωνία αυτή. Η ουσιαστική διαφορά, αν κατάλαβα καλά, ανάμεσα στην υπάρχουσα συμφωνία και τη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία είναι τονίζεται τη σημασία τη ευρύτερη κάλυψης σε πολιτικό, σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου που θα επηρεάσει ασφαλώς και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα και φαίνεται ότι συμφωνείτε με την ερμηνεία που έδωσα. Μήπως θα μπορούσατε να αναφέρετε, μας πείτε σύντομα τι σκέφτεται για πώς βλέπει τις ιδέες που ακούστηκαν εδώ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δεν είμαστε εκτελεστική εξουσία, είμαστε ένα κοινοβούλιο, αλλά χρειαζόμαστε, πρέπει να δούμε, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να δούμε αν αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα τα διάφορα θέματα. Τι λοιπόν θα μπορούσε κατά την άποψή σας να γίνει. Υπάρχουν κάποια προηγούμενα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω τις πληροφορίες που είχατε αναφέρει προηγουμένως ότι ξεκινούμε συνεργασία με το Κοινοβούλιο του Τουρκμενιστάν. Τους βοηθούμε να γίνουν ένα πραγματικό κοινοβούλιο, πραγματικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Επίσης, σε σχέση με τη θεσμική δομή, πιστεύω ότι έχουμε και την πρόβλεψη για αλληλεπίδραση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέσα στη σύνολη θεσμική διαδικασία. Αυτό σας δίνει λοιπόν και μια άλλη δυνατότητα συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη πρόταση της εισηγήτριας, το μόνο πράγμα για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή είναι να σας δίνουμε τακτικές εκθέσεις στην Υποεπιτροπή σας και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την κατάσταση στο Τουρκμενιστάν. Αν προβλέπετε πράγματι από το Κοινοβούλιο να υπάρξει ένας διαθεσμικός μηχανισμός, προφανώς θα πρέπει να τα μεταφέρω αυτά στους ανωτέρους μου, που είναι τώρα η Κομισιόν και στο μέλλον θα είναι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και προφανώς δεν μπορώ προσωπικά να εκφράρω γνώμη για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ λέει και η Πρόεδρος. Θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα αυτή την ιδέα και να έρθουμε και πάλι σε επαφή μαζί σα. Ίσως και είναι η στιγμή να κλείσουμε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι είναι ένα πιλωτικό κατά κάποιο τρόπο σχέδιο για να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες αρμοδιότητες του για τις διεθνείς συμφωνίες ώστε να αναλάβει πλήρως και σοβαρά τις ευθύνες και τις υποχρέωσεις του. Το εγχείρημα λοιπόν αυτό θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό ορόσημο είναι οι προθεσμίες για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στις 6 η ώρα στις 10 Νοεμβρίου θα εξεταστεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η δεύτερη εξέταση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία θα γίνει 25-26 Ιανουαρίου και θα έρθει στην Ολομέλεια το Μάρτιο του 2011. Αυτό είναι το αναθεωρημένο λοιπόν σχέδιο. Θα προσπαθήσουμε να το έχουμε στο μυαλό μας. Στις επερχόμενες εβδομάδες λοιπόν θα έχουμε και στενή συνεργασία με τους, ε, μεταξύ σκιωδών εισηγητών και της εισηγήτριας. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη, ευχαριστώ το Human Rights Watch, ε, το Open Society Institute, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τον εκπρόσωπο του ΙΠΑ του Επιτρόπου, του ΟΗΕ. Κλείνουμε αυτό το σημείο. Έχω να κάνω κάποιες αναγγελίες. Θέλω να καλωσορίσω τον ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Φιλιππίνες, εκπρόσωπο των εξαφανισμένων ή μάλλον ο ίδιος είχε εξαφανιστεί και επανήλθε. Θαυμάσιο νέο. Ε, η οργάνωσή του λέγεται Αντισαπαρεσίδο και ασχολείται με άτομα τα οποία έχουν απαχθεί στι Φιλιππίνες. Ο κ. Μαρέιμον Μανόλο ε, ήταν και ο ίδιο θύμα απαγωγή. παρέμεινε αγνοούμενο επί δύο χρόνια. Έχουμε την κυρία Κονσεψιόν Εμπένο, μητέρα ενός, μιας απειχθήσας κοπέλας, Κάρεν Εμπένο, που την απήγαν το 2006 στις κεντρικές Φιλιππίνες, η οποία όμως δεν έχει επανεμφανιστεί έκτοτε. Θα γίνει μία συνάντηση με τους φίλους μας από τις Φιλιππίνες σήμερα. Σας παρακαλώ, όσοι ασχολείστε με το Τουρκμενιστάν, ε, σημαντική συνάντηση, αλλά συνεχίστε έξω. Επομένως, θα γίνει από τις 4 παρατέταρτο μέχρι τις 5 παρατέταρτο στο δωμάτιο A3H1 ε, μια συνάντηση ε, για τις περιπτώσεις αυτές απαγωγών στις Φιλιππίνες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μας μιλήσετε για αυτό το πρόβλημα. Τώρα φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασης, αλλά έχουμε την συνάντηση του Διευρυμένου Προεδρίου. Μπορούμε να συνεχίσουμε αγγλικά και, με αγγλικά και γαλλικά μόνο με αυτές τις δύο γλώσσες. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή την διήμερη συνεδρίαση. Ακούσαμε πάρα πολλές πληροφορίες για το, την Τουρκία, το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και ασχοληθήκαμε με την ε, σημαντικότατη έκθεση, την ετήσια έκθεση της κυρίας Αντρικίενε. Η επόμενη συνάντησή μας η επόμενη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα γίνει στις 8 Νοεμβρίου. Γεια σας.